Colleagues, um, Ας ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Oh, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. 9 και 7 δηλαδή. Και έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Πάτρικ ε, Άιδεν από, τον, ε, από το Caesar προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων μαζί του. Βλέπω και ένα έδρανα εδώ. Παρόλο που πολλοί από εσά ζήτησαν να ενημερωθούν από το ΣΥΖΕΡ τι γίνεται. Οπότε, να ρωτήσω τους ε, πολιτικούς εδώ, τους συμβούλους και τα λοιπά, μήπως μπορούν να βρούνε τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές Εντάξει, καλή ποιότητα, αλλά και ποσότητα βοηθάει, αν είμαστε περισσότεροι. Η προσέλευση δεν είναι τόσο καλή. Όταν έχουμε να συζητήσουμε για κάτι τόσο σημαντικό όπως αυτό, θα έπρεπε να ήμασταν περισσότεροι παρόντες. Πάτρικ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα τάχτε φταίνε η τέφρα του ηφαιστείου που εμπόδισε του ευρωβουλευτέ να είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι, έχετε μια καλή δικαιολογία. Θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω λίγο για το που βρισκόμαστε όσον αφορά το ΣΥΖΑΡ και θα προσπαθήσω επίσης να μιλήσω και για το μέλλον, για την παρετέρω ανάπτυξη του ΣΥΖΑΡ που απαιτείται δράση από την Επιτροπή αυτή. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ να σας ενημερώσω για το Caesar. Τελευταία φορά που ήμουν εδώ σας εξήγησα την ιδιαίτερη φύση του προγράμματος Caesar, το κοινό εγχείρημα το οποίο έχουμε, στο οποίο συμμετέχει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε επεκτείνει την εταιρική μας σχέση με 13 επιπλέον εταίρους, έχοντας στο μυαλό μας δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να επεκτείνουμε την βάση μας των ε, παρόχων υπηρεσιών αεροπλοίες, ιδιαίτερα στο, στην Κεντρική Ευρώπη. Και το πετύχαμε. Έχουμε προσελκύσει την Πολωνία μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε όμως να δουλεύουμε. θέλουμε επίσης να έχουμε μαζί μας και άλλες χώρες που γυτνιάζουν με την Ευρώπη ή που έχουν ε, ιδιαίτερε σχέσει με την Ευρώπη, όπω είναι ο Καναδά ή το Μαρόκο. Ο δεύτερο στόχο που είχαμε υπόψη μα ήταν ότι θέλαμε περισσότερε μη ευρωπαϊκέ ε, βιομηχανίε, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε διαλειτουργικά τις τεχνολογίες του Caesar με άλλες περιοχές στον κόσμο. Η ιδέα ήταν ότι οι εταίροι αυτοί λειτουργούν ως σπόνσορες ιδιαίτερα σε αμερικανικές επιχειρήσεις και αμοιβαία υπάρχουν διακανονισμοί κατέρωθεν του Ατλαντικού. Ξέροντας ποιοι είναι οι περιορισμοί που υπάρχουν για τη συμμετοχή των Αμερικανικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα βάση του Next Gen. Έτσι λοιπόν έχουμε υπογράψει συμφωνίες με διάφορους χρήστες, με αρχές και έχουμε τώρα 200 εμπειρογνώμονες και 60 άτομα προσωπικό. Το Caesar είναι ένα από τα πιο περίπλοκα και φιλόδοξα προγράμματα στην Ευρώπη. Έχουμε 300 ε, προγράμματα, 16 πακέτα εργασίας, 110 επιχειρήσεις, 2.200 εμπειρογνώμονες που δουλεύουν και συνεργάζονται μαζί μας σε 23 διαφορετικές χώρες. Γι' αυτό και απαιτείται μεγάλη επένδυση σε προσπάθειες για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την αρχή της συνεργασίας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τους 2.000 εμπειρογνώμονες και τις διάφορες δυνατότητες διαχείρισης που δίνει το πρόγραμμα. Χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο από όσο αρχικά είχαμε προβλέψει, ομολογώ. Πετύχαμε όμως και καταφέραμε να το κάνουμε να δουλέψει. Και είμαι περήφανος που μπορώ σήμερα να σας πω ότι δύο χρόνια αφότου ξεκίνησε το πρόγραμμα έχουμε πετύχει να ξεκινήσουμε όλα τα επιμέρους προγράμματα και προχωράμε σε όλες τις τεχνικές δραστηριότητες ε, μέσα στον χρόνο που είχαμε προβλέψει και στα οικονομικά πλαίσια που είχαμε προβλέψει. Η πρώτη πρόκληση που είχαμε και σας το είπα και την προηγούμενη φορά ήταν να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν το πετύχαμε. Η επόμενη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα που έχουν νόημα. Και αυτή είναι μεγάλη πρόκληση γιατί 20 χρόνια τώρα κάπου 200 εκατομμύρια ευρώ είχαν επενδυθεί στην έρευνα έρευνα και επενδύσεις που έγιναν τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο από την Eurocontrol, αλλά χωρίς όμως πραγματικά αποτελέσματα που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό και αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε με τους εταίρους μας ότι όλα τα προϊόντα του Caesar θα πρέπει να έχουν δοκιμαστεί και επικυρωθεί μέσα σε ένα πραγματικά λειτουργικό περιβάλλον. Κατά το παρελθόν πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα είχαν δοκιμαστεί μέσα στα εργαστήρια και φαινόταν να μπορούν να αποδώσουν πραγματικά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τώρα όμως η προσέγγιση την οποία ακολουθούμε είναι ότι χρησιμοποιούμε λειτουργικά συστήματα με πραγματικές συνθήκες για να κυρώσουμε τα νέα εργαλεία και τις ε, διάφορες λειτουργικές διακασίες. Έτσι λοιπόν οι ελεκτές ενέργειες κυκλοφορίας, οι πιλότοι, οι μηχανικοί, όλοι αυτοί μπορούν να αξιολογήσουν κάτω από πραγματικές συνθήκες τα προϊόντα του ΣΥΖΕΡ. Η διεθνής ομάδα που βοηθάει σε αυτό μας βοηθάει και στην αξιολόγηση των ε, αλλαγών που γίνονται όσον αφορά την ασφάλεια και την απόδοση. Η βασική ιδέα είναι ότι εάν τα τεστ δοκιμής και επικύρωσης γίνονται ικανοποιητικά και έχουμε θετικά αποτελέσματα, τότε θα μπορούμε στη συνέχεια να τα εφαρμόσουμε και στην πράξη πολύ εύκολα. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα και απόφαση που πήραμε ήταν ότι αποφασίσαμε κάθε χρόνο να υποβάλουμε μία έκθεση απολογισμού του ΣΥΖΕΡ, η οποία αναφέρεται στα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη επικυρωθεί. Η πρώτη τέτοια έκθεση προβλέπεται ήδη για φέτο και θα συμπεριλαμβάνει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα όπως είναι η από απόσταση πύργη ελέγχου, χωρίς να έχουμε δηλαδή παρόντες τους ελεκτέ ενέργεια κυκλοφορία στα αεροδρόμια αυτά καθε αυτά. Πρόκειται επίσης για το συγχρονισμό των μέσων διαχείρισης ε, της άφηξης και της αναχώρησης για να έχουμε πιο μεγάλη απόδοση στα αεροδρόμια μας. Αποφασίσαμε επίσης να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά το αέρα, με 18 προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε. Πρόκειται δηλαδή για τους παρόχους υπηρεσιών ενέργειας κυκλοφορίας. Θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερες διαδρομές. Πρόκειται για τις διατλαντικές πτήσεις ως επιτοπλίστων όπου συνεργαζόμαστε εκεί με τους συναδέλφους μας από τις Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία και μπορούμε να καταλήξουμε σε εξοικονόμηση χρημάτων γιατί για παράδειγμα από 14, μάλλον από 1,4 τόνους καύσιμα από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση σε μια τέτοια διαδρομή. Ε, προσπαθούμε να δούμε το αντίστοιχο και για το Άμστερνταμ, τη Ζηρίχη, τη Βιέννη και τη Μαδρίτη. Χρηματοδοτούμε ως σπόνσορες 5.500 πράσινε πτήσεις επίσης, κάτι που έχει μεγάλη επιτυχία γιατί πολλέ αεροπορικές εταιρείε ζητούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμά μας. Τώρα λοιπόν δουλεύουμε με όλες αυτές τις ε, αεροπορικές εταιρείε και του φορεί, ώστε να έχουμε στην καθημερινότητά μα πια μόνο πράσινε πτήσει. Τώρα, πώς μπορεί να εφαρμοστεί το ΣΥΖΕΡ με συνεργασία τόσων διαφορετικών εταίρων που έχουν όμως έναν κοινό στόχο. Τι θα γίνει, πώς θα αναπτυχθεί παρετέρω το ΣΥΖΕΡ. Μόλις ολοκληρώσαμε μία μελέτη για τις επιπτώσεις του ΣΥΖΕΡ στην ευρωπαϊκή οικονομία. από μία ε, εξωτερική επιχείρηση έγινε η έρευνα αυτή. Ε, βοήθησε και την εταιρεία McKinsey Company. χρησιμοποίησαμε και πυρογνώμονε από τον ΟΣΑ, από τις χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξαμε τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Το ένα ήταν το business as usual, το δεύτερο ήταν να έχουμε ένα σχέδιο όπως προβλέπεται από το ΣΕΖΑΡ. Ένα τρίτο ήταν ο ένα συγχρονισμό της εφαρμογή του ΣΥΖΡ μεταξύ των διαφέρων ομάδων και το τέταρτο ήταν μια καθυστέρηση 10 ε, Μιλήσαμε για ένα ποσό μέχρι το 2030, 419 BR, που είναι 0,16% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και είναι το αντίστοιχο των 328.000 θέσεων απασχόλησης. Το σενάριο του αποσυγχρονισμού θα κατέληγε σε μια απώλεια ή στον διακεντρεύσιο 72.000 θέσεις απασχόλησης και με 10 χρόνια καθυστέρηση θα είχαμε απώλεια 189.000 θέσεων απασχόλησης. Μπορούμε εδώ να σχολιάσουμε, να πούμε ότι στη μελέτη αυτή αυτό που κοιτάξαμε ήταν τις άμεσες επιπτώσεις του ΣΥΖΑΡ στη, στον κλάδο. Δεν κοιτάξαμε τις έμεσες επιπτώσεις στον τουρισμό, για παράδειγμα, στις περιφερειακές οικονομίες κλπ. Η μελέτη λοιπόν δείχνει, και δεν μας εκπλήσει αυτό, ότι έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει συγχρονισμός. Και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με σωστό τρόπο, πώς μπορεί να λειτουργήσει καλά ο συγχρονισμός αυτός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει πάνω σε πρόταση για την ανάπτυξη του ΣΥΖΑΡ και από εκεί και πέρα θα αφήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσουν τη θέση του στο Κοινοβούλιο. Θέλω όμως να σας δώσω την προσωπική μου άποψη για αυτό που πιστεύω ότι αποτελούν τα δύο θεμέλια για την επιτυχή ανάπτυξη του ΣΥΖΑΡ. Πρώτον, πρέπει να έχουμε μια σωστή διακυβέρνηση. Η εμπειρία που έχουμε με τα διάφορα στάδια μέχρι τώρα δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει η συνεργασία, γιατί η δυναμική της ομάδας πολλές φορές βοηθάει πολύ περισσότερο από ότι ο τομικό ρυθμός του καθενός, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με δύσκολες αλλαγές. Ο θετικός ανταγωνισμός μέσα στην ομάδα βοηθάει να έχουμε τα καλύτερα δυνατόν παραδείγματα και να δουλέψουμε βάσει της αρχής αφού μπορούν οι άλλοι γιατί όχι εμείς. Και αυτό λέμε πολύ συχνά κι εμείς. Αφού μπορούν οι άλλοι ελεκτές γιατί όχι κι εμείς. Πάντως η αποκενού συνεργασία επιβάλλει κάποιους κανόνες και βασίζεται κύρια σε ένα σημείο αναφοράς, σε ένα άτομο δηλαδή, ο οποίος καλείται να πάρει αποφάσεις όταν αυτό χρειάζεται. Είναι πολύ βασικό αυτό για την ανάπτυξη του ΣΥΖΑΡ να υπάρχει μία ενιαία αρχή που θα λογοδοτεί όσον αφορά το πρόγραμμα και που θα μπορεί να πάρει αποφάσεις όταν οι επιμέρους ομάδες δεν μπορούν. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και αν το δούμε από τη διεθνή οπτική γωνία, γιατί η Κίνα, η Βραζιλία, η FAA έχουν μία ενιαία τέτοια αρχή το, η δεύτερη βάση, το δεύτερο θεμέλιο είναι η χρηματοδότηση του Σίζερ. Η αρχή του Σίζερ είναι να συμπεριλαμβάνει μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας όλους τους επιμέρους φορείς που ασχολούνται με τα διάφορα συστήματα διαχείρισης είτε είναι για τους ε, πύργους ελέγχου κυκλοφορίας είτε πρόκειται για άλλες λειτουργίες. Αυτά φαίνονται πολύ ωραία και εύκολα. Στην πράξη όμω, η ολοκλήρωση αυτή είναι ιδιαίτερα περίπλοκη τη δημιουργία εξαρτήσεις μεταξύ των επενδυτών ή των μετόχων που μερικές φορές έχουν αποκλίνοντα συμφέροντα. Για παράδειγμα θα σας φέρω το VHF radio ε, το οποίο σήμερα σημαίνει ο, κάτι για, τις για την επικοινωνία μάλλον μεταξύ αεροσκαφών και δάφους που χρησιμοποιεί η τεχνολογία του 1950 σήμερα ε, είναι απαρχιωμένο. Όμως δεν μπορούμε να το αφήσουμε παρά μόνο όταν όλοι έχουν τη νέα σύνδεση του διαδικτύου. Γι' αυτό οι αεροπορικές εταιρείες κοιτάνε η μία τι κάνει η άλλη. Περιμένουν να επενδύσουν οι άλλοι και όσο περνάει ο χρόνος φτηνένει και το προϊόν. Όμως ο εξοπλισμός θα έπρεπε να γίνει όταν όλα τα αεροσκάφη θα μπορούν να τον έχουν. Αλλά όπως σας είπα, ο καθένας κοιτά τι κάνει ο διπλανός του και κανείς δεν αποφασίζει να επενδύσει. Πάντως η ρύθμιση για τους ενιαίους εθέρες έχει ως στόχο μια τέτοια εφαρμογή, αλλά πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι κανόνες σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο και δεύτερον να υπάρχουν όρια που έχουν να κάνουν με το ότι περιμένει κανείς να εξοπλιστεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντως πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα από τα οποία αμοιβαία όλοι έχουν ε, να επωφεληθούν. Γι' αυτό και δουλεύουμε βάσει της αρχής best equipped, best served, ο καλύτερα εξοπλισμένος εξυπηρετείται και καλύτερα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αντιστάσεις, ιδιαίτερα από φορείς οι οποίοι φοβούνται ότι έτσι γίνεται πιο περίπλοκη δουλειά τους. Όσον αφορά τα οικονομικά κίνητρα, προσπαθούμε να βρούμε διάφορα οικονομικά μέσα, είτε πρόκειται για ομόλογα, είτε πρόκειται για δάνεια με χαμηλά επιτόκια κλπ τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε αν μη τι άλλο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία αλλαγή. Πάντω, οι περισσότερε από τι επενδύσει του ΣΥΖΑΡ θα γίνουν από τον κλάδο, από τη βιομηχανία, αλλά και ε, δημόσιο χρήμα μπορεί πολύ να βοηθήσει για την επιτυχία τη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Έτσι θα είμαστε περισσότερο ισχυροί και μπορούμε να αποφεληθούμε και από τη συνεκτική πολιτική του δημοσίου κάθε φορά. Τέλος θέλω να πω ότι το πρόγραμμα ΣΥΖΕΡ λειτουργεί καλά. Έγκαιρα, μέσα στο προβλεπόμενο κόστος και το 2011 έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αρχίσαμε να είμαστε και παρόντες στη διεθνή σκηνή με ένα μνημόνιο συνεργασία που υπογράφτηκε φέτο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ΗΠΑ που μα δίνει την εντολή να συντονίζουμε τι δραστηριότητε με του ε, εταίρου μα από τι ΗΠΑ. Δουλεύουμε και με την ΙΚΑΟ που είναι το Διεθνέ Συμβούλιο για την ενέργεια κυκλοφορία προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι δικές μας προδιαγραφές θα είναι και παγκόσμιες προδιαγραφές. Είναι πολύ βασικό η δουλειά αυτή να μην γίνει για το τίποτα, αλλά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία που συλλέγουμε εμείς για να αναπτυχθεί παρετέρω και το ΣΥΖΕΡ και να συνεχίσει να είναι όσο επιτυχές είναι και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πάτρικ. Υπάρχουν ορισμένοι ομιλητές εγγεγραμμένοι. Ο κύριος Ασάντα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη έκπληξη για μένα το ότι ομιλώ εξ του ΕΛΚ. Θα προσπαθήσω όμως να σας παρουσιάσω τη θέση μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Λυπάμαι που δεν έλαβα την παρουσίαση γραπτός. Θα το προτιμούσα για να είμαι καλύτερα προετοιμασμένος. Θα ήθελα να πω ε, εξ αρχής ότι είμαστε υπέρ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού, αυτού του σχεδίου, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου, του Σίζαρ, νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσει ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, γιατί αυτό θα σταθεί υπέρ της ενιαίας αγοράς. Όπως προγενέστερα χρησιμοποίησαμε και το σύστημα Galileo. Θα πρέπει να έχουμε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης των αερομεταφορών, ιδιαίτερα σε μικρότερα αεροδρόμια. Ε, δυστυχώς το σχέδιο Γαλιλαίο παρουσίασε μεγάλα προβλήματα. Εδώ στο Σίζαρ μιλάμε για ένα υψηλό κόστος διαχείρισης. Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε καθήκοντα τα οποία θα είναι ε, κερδοφόρα βραχυπρόθεσμα. Το πεδίο δραστηριότητας του ΣΥΖΑΡ είναι πολύ μεγάλο. Μιλάμε για εξοπλισμό αεροπλάνων, διαχείριση εναέριου χώρου, αερομεταφορές και ούτω καθεξής. Το θέμα του εξοπλισμού των αεροπλάνων είναι ύψης της σημασίας για την πολιτική αεροπορία και θα πρέπει να δούμε για ποιο εξοπλισμό μιλάμε στα αεροσκάφη. Υπάρχουν ε, αεροσκάφη τα οποία ε, δεν πληρούν τους όρους για παροχή νέων εξοπλισμών. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποιες είναι οι προαπαιτήσεις του ΣΥΖΑΡ, δηλαδή τι ραδιοσυχνότητες θα χρησιμοποιήσουμε στο σύστημα APSB. Επίσης, ως προς τη χρηματοδότηση ή τη συγχρηματοδότηση, έχετε κάποια συγκεκριμένη ιδέα. Αλκαντράουι. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Πατρίκη που ήρθε εδώ και μας έκανε αυτή την παρουσίαση. Είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ΣΥΖΕΡ και χαίρομαι που άκουσε ότι πάνε τα πράγματα καλά. Όμως σημασία έχει η φιλοδοξία που παρουσιάζει το πρόγραμμα αυτό και τα αποτελέσματα, αν είναι αντίστοιχα της φιλοδοξίας αυτής. Θα ήθελα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια αντίδραση για να ξέρω πότε θα ετοιμάσει την ε, δικιά της πρόταση για την παρετέρω ανάπτυξη του ΣΥΖΕΡ και πώς θα συνοδευτεί από πλευρά προϋπολογισμού το πρόγραμμα αυτό. Είναι καλό το ότι υπάρχουν και ιδιωτικέ επενδύσεις. Πάντως προβλέπετε, και αυτή είναι η ερώτηση, προβλέπετε μεσοπρόθεσμα επιπλέον ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Χρειάζεται ενθάρρυνση για να υπάρξουν περικοπές για παράδειγμα στα τέλη εναέριων κυκλοφοριών δεν ξέρω Πάντως από εσά αυτό που θέλω να ξέρω είναι να μου πείτε για σας το timing ποιο είναι όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην χαθεί χρόνος για σας και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στο πρόγραμμά σας. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε. Δεύτερον, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε παγκόσμιο επίπεδο, το Caesar δεν είναι ο μόνος παίκτη, έτσι, υπάρχει και το αντίστοιχο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι γίνεται με τη διαλειτουργικότητα, τι συμφωνία υπάρχει για τη διαλειτουργικότητα των διάφορων συστημάτων και τι γίνεται με την ε, πώληση προς τρίτες χώρες της ευρωπαϊκής αυτής τεχνολογίας. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Μπορούμε να βοηθήσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενδεχομένω ώστε το ΣΥΖΑΡ να μπορέσει να προσφέρει εκτός Ευρώπης. Κάτι ακόμα. Όσον αφορά την τέφαρα του ηφαιστείου, είναι επίκαιρο θέμα. Αναρωτιέμαι, σε τι βαθμό στο μέλλον θα μπορεί να βοηθήσει το ΣΥΖΕΡ ώστε να οριοθετηθούν καλύτερα οι απαγορευμένες περιοχές όταν έχουμε τέτοια, τέτοιες εκρήξεις ηφαιστείων με τέφρα. Μπορεί να γίνει αυτό. Τέλος, σε τι βαθμό το ΣΥΖΕΡ συμμετέχει στην ανάπτυξη των ενιαίων εθέρων. Ξέρετε ότι έχει μπλοκαριστεί κάπως το θέμα. Εσείς συμμετέχετε με το Σίζαρ. Νομίζετε ότι θα πάει καλά. Το 2012 θα τα έχουμε καταφέρει. Τι προβλέπετε. Και τώρα έρχομαι στο τελευταίο για τις επιπτώσεις στο κλίμα από το Σίζαρ. όντως μπορεί να βοηθήσει την προστασία του κλίματος. Είπατε 10% μείωση έχετε όσον αφορά τις εκπομπές. Ε, θα μείνετε σε αυτό. Και άλλη μια τελευταία ερώτηση, λέει Θέλω να μου πείτε για την συμπίεση, ξέρετε, στον αέρα. Υπάρχουν επιπτώσεις στο κλίμα. Αν υπάρχει καλή συνεργασία με τους μετεωρολόγους, ε, δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και με τις ε, αρχές ε, ελέγχου της κυκλοφορίας. Το ΣΥΖΑΡ συμμετέχει, πάει καλά μια τέτοια συνεργασία και τι δυνατότητες βελτίωσης υπάρχουν από τη συνεργασία αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον ομιλητή. Τέθηκαν ήδη ερωτήσει. Εγώ θα είμαι σύντομη και οφείλω να προσθέσω ότι αμέσως μετά πρέπει να αποχωρήσω από την αίθουσα. Ο συνάδελφός μου που κάθεται δίπλα μου θα με αντικαταστήσει. Τώρα, ερωτήσεις. Είπατε ότι πρόκειται και για το πράσινισμα εντό εισαγωγικών του αέρα, και ότι πρέπει να γίνει μια, ένα συντονισμός μεταξύ του ΣΕΣΑΡ και της προσπάθειας ανοιχτών εθέρων, ανοιχτών ουρανών. Η ερώτησή μου είναι Πού βρίσκεται η συνεργασία σας με τον κύριο Γιαρζεμπόσκι που είναι ο συντονιστής των ανοιχτών ουρανών από δικής μας πλευράς. Το άλλο που μας απασχολεί είναι βλέπετε την δυνατότητα με νέα περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας τα αεροσκάφη να είναι λιγότερο ευάλωτα, λιγότερο ευαίσθητα στην ύπαρξη σωματιδίων στον αέρα. Είπατε επίσης ότι χρειάζεστε την υποστήριξη της Ευρώπης. Εννοείται μονάχα χρηματοδοτικά, μονάχα λεφτά ή μπορούμε να προωθήσουμε το ΣΕΣΑΡ και με άλλο τρόπο με ανάληψη ε, ε, ε, διαφημιστικών ε, κινήσεων και ούτω καθεξής. Κύριε Φώστερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Πάτρικ για την ενημέρωση. Θα ήθελα να μας δώσετε και ένα αντίγραφο των διαφανειών που δείξατε. Το... Ήταν πάντως ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και κυρίως τώρα που επανήλθε το νέφος τέφρας. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο θα θυμάται και ο Μπράιαν Σίμψον πρόεδρος μας και ορισμένοι από τους παλαιότερους ευρωβουλευτές ότι είχαμε στηρίξει τότε την αλλαγή στην διαχείριση των εθέρων. Βεβαίως και είναι μακρά η διαδικασία αυτό που μας απογοητεύει κάπως τώρα είναι ότι οι χώρες μέλη δεν δεσμεύονται τόσο όσο θα έπρεπε. Βεβαίως και υπάρχουν πολλοί περιορισμοί οικονομικοί, δημοσιονομικοί και βεβαίως πρόκειται για χρήματα του δημοσίου τα οποία επενδύονται εδώ. Αλλά υπάρχει και ένας τεράστιος αριθμός εταιριών οι οποίες έχουν αναλάβει τη δέσμευση να επενδύσουν στην τεχνολογία που θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για τα προγράμματα αυτά Ανεξαρτήτως του τι θα προκύψει από την προσπάθεια αυτή, πρέπει να μείνουμε στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, διότι εντασσόμαστε σε παγκόσμια, διεθνή συστήματα και πρέπει να φροντίσουμε να κινούμαστε με τον ρυθμό και των υπολείπων. Και εμείς αλλά και οι συνάδελφοί μας της Επιτροφής Περιβάλλοντος γνωρίζουμε καλά ποιο είναι το κόστος τη συμφόρησης τους εθέρες και χρειαζόμαστε την προσπάθεια αυτή διότι υπάρχουν αρνητικοί αντίκτυποι και στην τιμή των εισιτηρίων. Και βεβαίως με την αύξηση της τιμής των καυσίμων τα πράγματα δεν βελτιώνονται. Ένας από τους συναδέλφους μας μίλησε για τα functional airspace blocks μέρος του SES e και έχουμε ακούσει και τον Γκέορκ ε, Γιαζεμπόφσκι ο οποίος τρέχει από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα και προσπαθεί να ενθαρρύνει την κίνηση προς τα εμπρός. Αλλά παρόλα αυτά η κίνηση είναι αργή. Πολλά λοιπόν πράγματα, πολλές πτυχές του θέματος που είναι και πολύ τεχνικές και περίπλοκες, δεν θα υπησέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μακροπρόθεσμα τα κέρδη είναι πολύ σημαντικότερα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε ακίνητοι. Θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Αλλά πάντως σας ευχαριστώ και πάλι Πάτρικ που προσήλθατε εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών και μας ενημερώσατε για το που βρίσκεστε. Όντως όμως χρειάζεται μια ισχυρή όθηση και νομίζω το αναγνωρίζουμε αυτό όλοι. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Καντσάν. Ευχαριστώ και Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς Πάτρικ. Θα ήταν χρήσιμο να είχαμε όντως τις διαφάνειες με κάποια μορφή. Θα μπορούσαμε, αν τις είχαμε λάβει και νωρίτερα, να προετοιμαστούμε καλύτερα για τη συζήτηση. Πάντως νομίζω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, ενιαίος Ευρωπαϊκό ουρανός. Στην ουσία το μέλλον υπαγορεύει την κίνηση αυτή. Και κυρίω μια ενιαία αρχή ασφαλεία Βρίσκω ότι είναι απαραίτητη. Και νομίζω ότι και αυτές οι κοινοπραξίες δημοσίου και ιδιωτικών φορέων είναι επίσης σημαντικές. Το ζήτημα της άμυνας απέναντι σε κυβέρνο επιθέσεις, σε τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ. Αυτά είναι επίσης ανισχυτικά. Είναι ανησυχητικά ανισχυτικά τα ενδεχόμενα αυτά. Θα ήθελα να μάθω την άποψή σας. Και δεύτερο ερώτημα, ποια συνεργασία προβλέπετε μεταξύ ΣΕΣΑΡ και χωρών της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Ρωσικής Κοινοπολιτείας. Μιλούμε για το ΝΑΤΟ, μιλούμε για άμυνα. Το ΝΑΤΟ έχει και το σκέλος του στρατιωτικού το στρατιωτικό μάλλον σκέλος ε, της, ε, του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και μπορεί να συμβάλλει στην βελτιστοποίηση των ε, ροών. Η σχέση και με την επόμενη γενιά τεχνολογία είναι σημαντική. Ολόκληρη η αμερικανική βιομηχανία είναι το ερώτημα προς τα που θα κατευθυνθεί. Για να είναι συμβατά τα συστήματα. Θα ήθελα να μιλήσω για την σχέση μεταξύ ΣΕΣΑΡ και ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Αυτή η συνεργασία πώς επηρεάζει την απόδοση όταν μιλούμε για λειτουργικά air block. Και έχω και άλλη μια ερώτηση. Ποια είναι τα προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια ή την χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε ότι συμμετέχουν στην κοινή αυτή πρωτοβουλία και χώρες, μέλη, αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Και είναι σημαντικό νομίζω να γνωρίζουμε εάν θεωρείτε ότι υπάρχει ανεπαρκής χρηματοδότηση και ποιες δυνατότητες βλέπετε για να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό. Εν τέλει, μια ακόμη ερώτηση, εάν δηλαδή η κοινή πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό και κατασκευή νέων μηχανών που θα ρηπαίνουν λιγότερο, θα είναι πιο αποδοτικές από άποψη κατανάλωσης ενέργειας, εάν αυτή η εξέλιξη θα λάβει υπόψη και την παρούσα κατάσταση, δηλαδή το νέφος τέφρας, αλλά επίσης και ανεμοθίελες, ή αμμοθίελες μάλλον, αμμοθίελες, δηλαδή ε, νέφη άμμου. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα σήμερα το πρωί. Πάντα η Επιτροπή μας θέλει να συζητάει και να στηρίζει στις χρηματοδομικές προοπτικές το έργο σας. Την βελτίωση του Ευρωπαϊκού Ενέργειου Χώρου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τώρα που χρειαζόμαστε ενίσχυση του χώρου αυτού και θέλουμε να στηρίξουμε την τεχνολογία, την βιομηχανία, το ΣΥΖΑ, Ξέρουμε ότι έχει μεγάλη σημασία και για το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας δώσετε και τέτοια στοιχεία. Για παράδειγμα, ένα βασικό στοιχείο είναι το κατά πόσο από το ΣΥΖΑΡ, όχι μόνο Eurocontrol, που είναι ο συνομιλητής του ΣΥΖΑΡ, αλλά μήπως θα μπορούσατε να βοηθήσετε με το ζήτημα του νεφουστέφρας. Τι μπορεί να κάνει το ΣΥΖΑΡ είτε τώρα είτε στο μέλλον για να ξέρουμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Caesar για να αντιμετωπίσουμε και τέτοια προβλήματα όπως είναι αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Και από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να τονίσω, Πάτρικ, τα θέματα που έθιξαν ε, η πολιτική μας ως προς την διασύνδεση του Σίζαρ και του ενιαίου ουρανού και την εργασία του κυρίου Γιαρζεμπόφσκι επί του θέματος. Θα πρέπει να αποστείλουμε σαφή μηνύματα για το τι θα ήταν χρήσιμο και τι όχι. Επίσης, ε, μας απασχολεί και ένα άλλο θέμα ως προς το πώς προχωρούμε με τα κράτη-μέλη. Μας ανησυχεί, γιατί όπως είπε η κυρία Φώστερ, δεν πρόκειται για ένα νεογέννητο, πρόκειται για ένα παιδί που ήδη φτάνει στην ηλικία της εφηβείας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που βρίσκεται σε εμβριακή μορφή. Είναι ένα σχέδιο που έχει προχωρήσει αρκετά και μέχρι το 2011 περιμέναμε κάποιες εξελίξεις. Με ενδιαφέρει η διασύνδεση με το θέμα του ενιαίου ουρανού και ιδιαίτερα όταν εκρήγνεται ένα ηφαίστειο τα κράτη-μέλη λένε ότι πρέπει να προωθήσουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Όταν όμως δεν υπάρχουν εκρήξεις, δεν ασχολούνται τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα. Ίσως χρειαζόμαστε περισσότερες εκρήξεις έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν σοβαρότερα με το θέμα. Επίσης, η έρευνα McKinsey, στην οποία αναφερθήκατε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα τα σενάρια περί ευεργετημάτων του Σίζαρ. Γιατί ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι η ανησυχία, η αμφιβολία που, έχουν και ορισμένοι, που εκφράζουν και ορισμένοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ότι αυτό το σχέδιο απειλεί την εργασία τους. Αποτελεί απειλή για τις θέσεις εργασίας και από ό,τι φαίνεται από την έρευνα McKinsey δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εάν λοιπόν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, πώς μπορούμε να πείσουμε τους ελεγκτές αέριας κυκλοφορίες και ιδιαίτερα τους Γάλλους ελεγκτές ότι αυτό είναι μια πραγματική ευκαιρία. Δεν είναι απειλή. Δεν αποτελεί απειλή για την εργασία τους που δεν αφορά μόνο τους Γάλλους ελεγκτές, εκφράζεται γενικότερα ο φόβος ότι ε, τίθενται εν κινδύνο θέσεις εργασίας, θέσεις απασχόλησης. Άρα πώς μπορούμε να πείσουμε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι αυτό θα ήταν κάτι το θετικό. Δεν ξέρω κατά πόσο η Επιτροπή θέλει το λόγο, κύριος Μπόλτου. Πρόεδρε, ε, δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται. Θα απαντήσω στα κεντρικά ζητήματα πρώτα. Ε, Μάθιου, ε, θέλεις να ακούσει την απάντηση του Πάτρικ, μήπως πει κάτι λάθος να τον διορθώσεις. Ε, Πάτρικ, θέλεις καταρχήν να απαντήσεις και μετά θα λάβει το λόγο η Κομισιόν. Μπράιαν, πολλά ε, θέματα εθίγησαν και θα προσπαθήσω να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Σχέση, συσχετισμό Σίζαρ και ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Το Σίζαρ ε, εντάσσεται στο ενιαίο σχέδιο, δηλαδή ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το Σίζαρ και Τούμπαλιν. Όταν μίλησα λοιπόν για τις νέες τεχνολογίες, για τον νέο εξοπλισμό, ήθελα να πω ότι η νομοθεσία θα μας βοηθήσει να ε, εφαρμόσουμε ώστε να ισχύσει δηλαδή αυτός ο, ε, εξοπλισμός και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον ίδιο τύπο τεχνολογίας που μπορεί να γίνει μέσω ενιαίου ε, ουρανού. Συναντήθηκα με τον κύριο Ζεμπόφσκι και θα πρέπει να πω ότι τα φάμπη οικοδομήθηκαν εντελώς ε, μάλλον ετεροχρονισμένα σε σχέση με την εφαρμογή του ΣΥΖΑΡ. Δεν έγινε πραγματική συζήτηση μεταξύ των λειτουργικών ΦΑΜΠ και του Σίζαρ. Μιλούσαμε για διαθεσμικές, διαθεσμικές συμφωνίες μέσα στα πλαίσια των σχεδίων άμυνας και μιλούσαμε μόνο για τον εναέριο ε, χώρο και τις υποδομές που χρειάζονται. Πρόκειται για βραχυπρόθεσμους στόχους για να έχουμε ε, γρήγορη κερδοφορία και ε, δεν έγινε λόγος για νέες τεχνολογίες τότε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε καλύτερα αυτά τα σχέδια με βάση νέα συστήματα. Όμως δεν υπάρχει ούτε ένα φαμπ που να έχει το ίδιο σύστημα. Όλα τα functional airspace blocks έχουν διαφορετικά συστήματα και γι' αυτό περιμένουμε έτσι ώστε το ΣΥΖΑΡ να είναι αρκετά όριμο για να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Αρχίσαμε λοιπόν με τα FAB, με μερικά από αυτά τα μπλοκ, όχι όλα, μέσα στα πλαίσια του διαθεσμικού ε, διαλόγου και δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία. Αλλά αρχίσαμε τις ε, συζητήσεις με την Ιλλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να δούμε πώς αυτά τα μπλοκ του εναέριου χώρου, τα λειτουργικά μπλοκ μπορούν να λειτουργήσουν. Και πώς με ένα νέο σύστημα, εάν υπάρξει νέο σύστημα, δεν θα πρέπει να συντονιστούμε με κάθε ε, κράτος ξεχωριστά ή με κάθε εναέριο χώρο, κρατικό εναέριο χώρο, αλλά με το λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου. Ως προς το ηφαίστειο την τέφρα δεν μπορεί να υπάρχει προβλεψιμότητα με βάση τα παρόντα συστήματα. Θα μπορούσα να σας πω λοιπόν, θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να σας πω ότι όλα επιλύονται με το Σίζαρ, ότι είναι πανάκια, αλλά δεν είναι. Ο Μάθιου θα σας πει ότι πρόκειται για μία διαδικασία λήψης αποφάσεων, δηλαδή ποιος αποφασίζει και ποιος λογοδοτεί. Επ' αυτού το Caesar είναι απλώς τεχνολογία, ένα μέρος της τεχνολογίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε καλύτερους τρόπους για την διάδοση πληροφοριών στους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και δεύτερον να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε έναν ακριβέστερο τρόπο επιβολής ε, δεσμεύσεων και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε έκτακτες καταστάσεις όπως η φεστιακή τέφρα. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιστοποιήσουμε την αντιμετώπιση αυτών των έκτακτων καταστάσεων. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει η χνηλάτιση της τέφρας ή κάτι τέτοιο ως προς τη συνεργασία με τις άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Υπάρχουν σήμερα δύο βασικά πρόγραμμα, το ΣΥΖΑΡ και το Ιαπωνικό σύστημα, το σύστημα των ΙΠΑ. Και οι Ιάπωνες προσπαθούν ε, να προωθήσουν ένα σύστημα, αλλά δεν είναι ακόμα λειτουργικό. Η συνεργασία μας με τις ΙΠΑ είναι πολύ καλή και έχουμε μια σωστή ε, και επαρκή τεχνική συνεργασία για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Βεβαίως θα ανακύψουν ζητήματα και πάλι. Δηλαδή υφίσταται ανταγωνισμός ε, των βιομηχανιών μέσα στα πλαίσια του ΣΥΖΑΡ και των ΙΠΑ. Και θα έχουμε και συγκρουόμενα ε, συμφέροντα ως προς τις προδιαγραφές ή τα χρονοδιαγράμματά μας. Θα πρέπει λοιπόν να βρίσκεται σε καλή θέση η Ευρώπη για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν οι μηχανισμοί για να συζητήσουμε με τους Αμερικανούς το όλο θέμα και να επιλύσουμε τα ζητήματα που ανακύπτουν. Δεν βρισκόμαστε σε απόλυτο αλλά σχετικό ανταγωνισμό. Το οικονομικό κλίμα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν δύο πρότυπα, θα υπάρχει ένα διαλειτουργικό πρότυπο και θα υπάρχει ανταγωνισμός στη βιομηχανία ως προς τα, ε, τις πατέντες, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ούτω καθεξής. Μπορούμε όμως να το συζητήσουμε με τους Αμερικανούς. Ή θα συμφωνήσουμε σε κάτι ή θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και τότε θα τεθεί σε άλλα επίπεδα η συζήτηση στο ΙΚΑΟ έχουμε αρχίσει τις συζητήσεις με ορισμένες χώρες, με τη Λατινική Αμερική, επί παραδείγματι. Συνεργαζόμαστε και με το Μεξικό και τη Βραζιλία, έτσι ώστε τουλάχιστον να γνωρίζουμε για το τι γίνεται και ποια είναι τα σχέδιά μας και τα σχέδιά τους. Αυτό αφορά το Μεξικό και τη Βραζιλία. Προσπαθούμε να συντονίσουμε τα χρονοδιαγράμματά μας και τις δραστηριότητες όταν πρόκειται για εξοπλισμό αεροσκαφών. Δεν υπάρχει εξοπλισμός που είναι ασύμβατος για τα αεροσκάφη που πρέπει να μπουν στον εναέριο χώρο της Λατινικής Αμερικής. Συζητούμε και με την Κίνα και την Ινδία και θα πρέπει να πω ότι έχουμε κάπως καθυστερήσει σε σχέση με τις ΙΠΑ. Υπάρχουν ε, μνημόνια ε, συνεννόησης με την Ιαπωνία, Αυστραλία, Καναδά και ούτω καθεξής, αλλά αυτό που προσπαθούμε είναι να εξασφαλίσουμε ώστε να υπάρχουν κοινά χρονοδιαγράμματα για να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσει, οι προαπαιτήσει σε όλες τις περιφέρειες. Αυτό που έχει σημασία είναι τι θα κάνει ο ΙΚΑΟ, διότι ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Πολιτικής Αεροπλοείας είναι αυτός που αποφασίζει τα παγκόσμια πρότυπα και έχει σημασία τι θα αποφασίσει ο ΙΚΑΟ θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν παρόντες στις ε, τεχνικές ε, επιτροπές του ΙΚΑΟ έτσι ώστε να εισακουστεί η δική μας φωνή ως προς τον ε, έλεγχο ενέργειας κυκλοφορίας και τη, τη μετεωρολογία και τις κλιματικές αλλαγές θα ήθελα να πω ότι το ΣΥΖΑΡ θα έχει επιπτώσεις, θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον γιατί στόχος είναι να έχουμε 10% χαμηλότερες εκπομπές αναπτύσσει. Άρα είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να φτάσουμε ήδη στο 3 με 4% μείωση εκπομπών αναπτύσσει. Υπάρχουν λοιπόν, ε, υπάρχει δυνατότητα να φτάσουμε αυτό το 10%. Αυτό σημαίνει ότι μέσω του ΣΥΖΑΡ μπορούμε να φτάσουμε σε σχέδια τα οποία θα μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θα φτάσουμε σε μια κατάσταση ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές. Το ίδιο ισχύει και με το πρόγραμμα των ΙΠΑ. Στο ΣΥΖΑΡ όμως δεν εργαζόμαστε ε, για να δούμε ποια είναι η επίπτωση της αεροπλοείας στη συνολική, στις συνολικές κλιματικές αλλαγές. Δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις και εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται έρευνα για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις επί, των, επί της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Δεν έχουμε την τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο. Όμως ε, συνεργαζόμαστε με τις αρχές της μετεωρολογίας, συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να είναι και εκείνοι οι φορείς ε, κοινωνή της εργασίας μας και να λάβουμε τα πρότυπα μετεωρολογίας για τον τρόπο οικοδόμησης των δικών μας συστημάτων. Αν λοιπόν σε κάποιο στάδιο δούμε ότι υπάρχουν ε, περιορισμοί, μπορούμε στο ΣΥΖΑΡ να διαχειριστούμε πολύ καλύτερα αυτούς τους περιορισμούς. Ε, ε, ως προς τη γρήγορη κερδοφορία προσπαθούμε να συνεργαστούμε για, τις, για τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, για τέτοια σχέδια και όπως σας είπα για τους απομακρυσμένους πύργους ελέγχου αυτό θα μπορούσε, το σχέδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί από του χρόνου. Και έτσι θα υπήρχαν ε, σοβαρές επιπτώσεις ως προς την αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα στη Βόρεια και Νότια Ευρώπη, όπου υπάρχουν αεροδρόμια όπου οι ελεγκτές ελέγχουν πέντε αεροσκάφη την ημέρα. Οι ίδιοι ελεγκτές θα μπορούσαν να ελέγχουν πέντε αεροδρόμια ημερησίω. άρα να είναι πιο αποτελεσματικό το σχέδιο. Άρα επανέρχομαι σε ένα από τα σημεία που φίξατε Τι θα γίνει με το εργατικό δυναμικό των ελεκτών, διότι η απομακρυσμένη πύργη σημαίνει ότι θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις επί της εργασίας. Όμως θα υπάρχει καταρχήν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση γιατί ένας ελεγκτής που ελέγχει μόνο πέντε αεροσκάφη ημερησίως, μην μου πείτε ότι είναι ικανοποιημένο από την εργασία του. Επίσης, εμείς συνεργαζόμαστε με τα συνδικάτα για να δούμε πόσο νέος εξοπλισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, να υπάρχει λιγότερο στρες, λιγότερη κόποση και ούτω καθεξής. Αυτός ο εξοπλισμός θα τους ε, βοηθήσει να έχουν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Άρα στα πλαίσια του Caesar θα μπορούσαμε να έχουμε ε, ένα, την αντιμετώπιση περισσότερου ε, φόρτου εργασίας με τους ίδιους ελεγκτές. Θα υπάρχει κέρδος δηλαδή, διότι ο ίδιος αριθμός ελεγκτών θα έχει το διπλό φόρτο. και νομίζω ότι μέχρι τούδε το σχέδιο προχωρά αρκετά καλά. Ως προς το ρόλο των κρατών μελών και την ε, υποστήριξη του Κοινοβουλίου, την ενδεχόμενη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εργαζόμαστε σε μια συντηρητική βιομηχανία. Οποιαδήποτε αλλαγή είναι πολύ δύσκολη. Στο ΣΥΖΑΡ όπως και στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μπορώ να σας πω ότι τα κράτη-μέλη ε, κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά μετά παλινοδούν. Θα ήθελα λοιπόν να μας βοηθήσετε, διότι όταν μιλάμε για εφαρμογή τεχνολογικών σχημάτων, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ε, αμφισβήτηση από πολλούς φορείς διότι δεν υπάρχουν ε, άμεσα αποτελέσματα. Αλλά μακροπρόθεσμα τα κέρδη είναι μεγάλα για ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό ο ευρωπαϊκός χώρος μας υπηρετεί, αλλά αν δεν ασκήσει πίεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση στα κράτη-μέλη, θα αντιμετωπίσουμε ορισμένες δυσκολίες. Οι εδώ έχουν ένα μείζον πλεονέκτημα έναντι ημών. Δηλαδή υπάρχει ένα κράτος. Και όταν πιστεί, πίστηκε. Ενώ εδώ μπορείτε να έχετε ένα που συμφωνεί, αλλά δεν αρκεί αυτό για την εφαρμογή του σχεδίου. Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά προσκόμματα για την εφαρμογή του ΣΥΖΑΡ. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε και για ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών. Στο Σίζαρ θέλουμε να έχουμε προτεργάτες, νικητές, ας το πούμε έτσι, ως προς τους απομακρυσμένους πύργους ελέγχου, οι Σουηδοί είναι αρκετά θαραλέοι και προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο. Όταν το εντάξαμε στο πρόγραμμα εργασίας, κανένας άλλος εκτός από τους Σουηδούς δεν δέχτηκε να συνεργαστεί. Τώρα όμως που βρισκόμαστε στο στάδιο δοκιμών και βλέπουμε ότι υπάρχει τεχνολογία και οι ελεγκτές είναι ε, αρκετά ικανοποιημένοι, βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες που μας λένε ότι δεν θέλω τυπικά να συμμετέχω, αλλά με ενδιαφέρει πολύ αυτή η εργασία άτυπα. Άρα μπορούμε να προωθήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών για να επιταχύνουμε την εφαρμογή του ΣΥΖΑΡ, αλλά θα χρειαστούμε μεγάλη υποστήριξη και από εσάς για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ελπίζω να κάλυψα όλες τις ερωτήσεις. Ως προς το θέμα της άμυνας, και εμείς ανησυχούμε για την ευαλωτότητα του συστήματος αυτού. Γι' αυτό αρχίσαμε τις συζητήσεις με τις αρχές άμυνας, ιδιαίτερα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και τον ΝΑΤΟ, για να επιτελεστούν στόχοι ασφάλειας του ΣΥΖΑΡ και πριν από το τέλος του έτους θα ορίσουμε τις ενδεχόμενες απειλές για να υπάρχει η σωστή διασφάλιση και για να μην διατρέχουμε κινδύνους μέσα στο, στα πλαίσια του συστήματος Caesar. Νομίζω ότι τα, νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Κύριε Μπόλτουιν, τώρα μπορείτε να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ να λάβω το λόγο. Ευχαριστώ που οργανώσατε τη σημαντική αυτή ακρόαση. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που μπορέσαμε να εμπαθύνουμε στα θέματα αυτά. Δεν θα σας ψυχαγωγήσω βέβαια πολύ. Θα προσπαθήσω πρώτα, να, θα πω μόνο πρώτα ότι υποστηρίζω τα όσα είπε ο Πάτρικ Κι και απάντησε στις ερωτήσεις σας. Αυτό που είπε στην αρχή για τον ομφάλιο λόρο μεταξύ του του ε, ε, Ενίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και του προγράμματο ΣΕΣΑΡ είναι σωστά και γι' αυτό ευχαριστώ τον Πατρική για την πραγματική, πραγματικά η ε, ηγετική του ε, ικανότητα και, και διάθεση στο θέμα αυτό. Αυτό που έχει προσφέρει το πρόγραμμα είναι η συλλογή πολλών και σημαντικών δυνάμεων, δεξιοτεχνιών του, και καινοτομία του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και την ε, ισχύ του δημόσιου τομέα. Όλα τα πλεονεκτήματα, τα ωφέλη για τη βιομηχανία, για τον εναέριο έλεγχο, για τους επιβάτες είναι πραγματικά. Και η μακροοικονομική μελέτη στην οποία αναφέρθηκε ο Πάτρικ θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και νομίζω θα εξηγήσει σε μεγάλο βαθμό και, τη, και τα οικονομικά θεμέλια αλλά και τους λόγους για τους οποίους αξίζει να υποστηρίξουμε το, το σύστημα. Τώρα θεωρώ ότι μπαίνουμε σε δύσκολα νερά καθώς προχωρούμε προς την εφαρμογή του συστήματος. Εσείς κύριε Χαντράουι θέσατε μερικές κέρυες ερωτήσεις για το πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα διαχειριστούμε τον προϋπολογισμό και πώς μπορούμε να αποφύγουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Αν μου επιτρέπετε λίγα λόγια για καθένα από τα ε, σημεία αυτά. Όπως είπε ο Πάτρικ Κι, πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για όλους τους ενδιαφερομένους για να εφαρμόσουν τις τεχνολογίες αυτές με τρόπο συγχρονισμένο και συντονισμένο. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα, τα διαθέσιμα μέσα για να προχωρήσουμε για τον ανοιχτό ουρανό. Αυτό που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να κάνουμε μια high-level task force με προσώπους... Ε, του ε- Eurocontrol, τον Μακμπίλαν, τον Πάτρικ από το ΣΕΣΑ και άλλους οργανισμούς υπό ε, την αιγίδα του Ματιού Ρίτς ε, που ήταν εχθές μαζί σας και αυτή η τετραμελής επιτροπή τώρα θα συντάξει έκθεση η οποία θα καταλήξει στον αντιπρόεδρο κύριο Κάλλας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε ήδη μέσα στο τρέχον έτος να έχουμε να, ε, φέτος ήδη να υπάρχει, το, το σχετικό έγγραφο που βάζει επιτροπή Δεν μπορώ να πω πιο, ε, με μεγαλύτερη ακρίβεια ε, χρονοδιάγραμμα. Και ε, θα δείτε από το αρχικό έγγραφο του Δεκέμβρη ότι έχουμε εκεί περιγράψει διαφορετικά σενάρια τα απορίσματα της ε, Task Force είναι ότι κανένας από τους παράγοντες μόνος του δεν μπορεί να αποδώσει αυτή την ε, ορθή διαχείριση. Γιατί γι' αυτό χρειάζεται το πολιτικό επίπεδο, το προγραμματικό επίπεδο και το επίπεδο τέλος του έργου. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε, συντονισμό των τριών επίπεδων. Είναι δύσκολο και είναι δύσκολο και από πλευρά concept να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε αυτό το μείγμα των κινητήριων δυνάμεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και πιο συγκεκριμένα τώρα για τη χρηματοδότηση. Έχουμε εντοπίσει ορισμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορου τρόπου, σε συνδυασμό βεβαίω και με τα απαραίτητα κίνητρα, ώστε να διασφαλιστεί αυτό ο συγχρονισμό. Για την ώρα δεν βλέπουμε να υπάρχει ανάγκη ειδικών μηχανισμών χρηματοδότησης του ΣΕΣΑΡ. Είναι σαφές όμως, πολύ σαφές και επιθυμώ να εγγραφεί και στα πρακτικά, ότι θεωρούμε ότι θα χρειαστεί χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Φώστερ δικαίω το επεσήμανε. Γνωρίζουμε βεβαίω ότι οι ε, συνθήκες από άποψη δημοσιονομική είναι δύσκολοι για τις χώρες μέλη, είναι δύσκολε μάλλον, αλλά δεν βλέπω να προχωρεί το έργο χωρί ε, χρηματοδότηση της Ένωσης. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν προχωρώ σε εικασίες, αλλά ε, περίπου 30 δις ευρώ θα χρειαστεί θα χρειαστούν για την φάση της εφαρμογής. Και ρεαλιστικά πολλοί μιλούν για 10% συμβολή πόρων ε, κοινοτικών. Βέβαια, μπαίνουμε τώρα ούτως ή άλλως ε, στην περίοδο της ε, νέας δημοσιονομικής πρόπτικης και θα γνωρίζουμε περισσότερο και πόσα χρήματα θα χρειαστούν αλλά και πόσα θα είναι διαθέσιμα. Ένα τελικό σχόλιο για τα λεγόμενα FAB functional airspace blocks. Δεν θα πω πολύ περισσότερα από τα όσα είπε ο Πατρικίδη ότι τα έχουμε ήδη συζητήσει αυτά τα πράγματα εδώ στην Επιτροπή σας και με τον κύριο Γιαζεμπόσκη. Εγώ επιθυμώ εδώ και δημοσία να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαζεμπόσκη για την δέσμευσή του, για την δουλειά που έχει κάνει αλλά καθώ και την Επιτροπή Μεταφορών. Δεν είναι εύκολε οι υποθέσει αυτέ, είναι όμω πάρα πολύ σημαντικέ. Έχουν σχέση με θεσμικά ζητήματα και μέσα στι χώρε μέλη, αλλά και ανάμεσα στι χώρε μέλη. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Η προθεσμία του Δεκεμβρίου 2012 είναι πραγματική. Ορισμένοι θεωρούν ότι α, καλά δεν πειράζει μέχρι τότε έχουμε καιρό. Δεν έχουμε, διότι οι αλλαγές είναι δύσκολο να επιβληθούν. Γι' αυτό ο Αντιπρόεδρος Κάλλας επιθυμεί να δει πραγματική αλλαγή, να προχωρεί και στο θέμα των ΦΑΜΠ. Και η πίεση εξακολουθεί, όπως είπα, να ασκείται. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που διοργανώσατε την παρούσα ακρόαση. Μιλήσατε και για την ηφαιστειακή τέφρα προηγουμένω. Πολύ ευχαρίστω να επανέλθω μετά. Στα διάφορα, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσά, Πάτρικ. αν μπορείτε να μας δώσετε ένα αντίγραφο των διαφανειών σας για να διανύμουμε στα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και τέλος πώς είναι δυνατόν τα ταξί των Βρυξελών να βρίσκονται στην πρωτοπορία της χρήσης των ε, υψηλών συχνοτήτων των VHF δηλαδή, αλλά σίγουρα πάντως δεν είναι μπροστά σε άλλα θέματα τα ταξί των Βρυξελών. Uh, Ανταλλαγή απόψεων για την επιτροπολογία για τις άδειες χειριστών. Ίσως καλά είναι να αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά ο κ. Αλχατράουι ως διαρκής εισηγητής. Θέλετε να κάνετε πρώτα μια σύντομη εισαγωγή κύριε Χατράουι. Καλά λοιπόν, τότε να πετάξω τις σημειώσεις του Πρόεδρου αφού μου λένε άλλα πράγματα. Σύντομη εισαγωγή λοιπόν. Ευχαριστώ. Ήθελα το λόγο για να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες να συμπεριλάβει στην παρουσίασή της στη συνέχεια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Ήρθαμε να ακούσουμε και να καταλάβουμε πώς προχωράει αυτή η υπόθεση. Έχουμε ερωτήσεις προς το Συμβούλιο. Οι συντονιστές μεταξύ μας αποφασίσαμε στην επόμενη συνεδρίαση συντονιστών να αποφασίσουμε τελικά κατά πόσο οι διαδικασίες είναι σύμφωνες ή θα πρέπει να έχουμε ένα ψήφισμα. Πάντως, Καταρχήν, είμαστε υπέρ ενό ευρωπαϊκού συστήματο ε, αδειών για του πιλότους μα. Είναι κάτι που συνάδει με τι εξελίξει στην αγορά. Έχω όμω τρει ερωτήσει. για πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε ακόμα αρκετά καλά. Πρώτον, το cruise relief είναι εξ αποστάσεως πτήσης, είναι κατά κάποιο τρόπο η οδήγηση του αεροπλάνου με cruise control. όπου διάφοροι συνπιλότοι με λιγότερα προσόντα ε, μπορούν να αποτελέσουν πλήρωμα ενό του σκάφους. Οπότε υπάρχει ο φόβος μήπως με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε δύο κατηγοριών συνπιλότους. Συνκυβερνήτες, πιο σωστά. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε περισσότερα πράγματα από αυτού. Δεύτερον, πολύ συχνά τελευταία ακούμε για πιλότους, κυβερνήτες από ιδιωτικά, ιδιωτικές εταιρείες οι οποίοι εμπλέκονται στο σύστημα αυτό. Όσο δεν υπάρχει συμφωνία για αναγνώριση ε, αμοιβαία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, χρειάζονται οι κυβερνήτες αυτοί δύο άδειες, Κάτι το οποίο κοστίζει παραπάνω χρήματα. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Τι γίνεται με την αμοιβαία αναγνώριση λοιπόν μεταξύ Πολιτειών και Ευρώπης. Και τέλος, ιδιαίτερα τους συναδέλφους ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο αφορά αυτό το θέμα του νέφους και των ε, νεφών γενικότερα που πιο συχνά έχουμε εκεί. Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα όταν υπάρχει χαμηλή ορατότητα. Πώς μπορούν τα αεροσκάφη να το ξεπεράσουν αυτό, τι δυνατότητες έχουν. Αυτές τις τρεις ερωτήσεις είχα και ελπίζω στην παρουσίασή σας να μας απαντήσετε σε αυτές. Ευχαριστώ. Καλώς, λέει Πρόεδρος, κύριε Μπόλτουιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Ολκάντραουι που με τέτοια σαφήνεια έθεσε τις ερωτήσεις του. Όντως θα προσπαθήσω να τις απαντήσω. Μου ζητήσατε έτσι και να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Όπως γνωρίζετε, ο κανονισμός 216 του 2008 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάζει καινούς κανόνες στον τομέα της ε, αεροπλοίας και δίνει ένα ρόλο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ασφάλειας ενέργειας κυκλοφορίας. Συμπεριλαμβάνονται εκεί και κανόνες όσον αφορά τις άδειες των κυβερνητών των αεροσκαφών. Κάτι άλλο που λέει ο κανονισμός λέει ότι οι κανόνες αυτοί ισχύουν από τις 8 Απριλίου του 2012. Αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί του συστήματος. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ συγκεκριμένη προθεσμία για όλους μας. Όπως είπα πριν, από λίγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη βοήθεια της Υπηρεσίας ε, Ασφάλειας και Κυκλοφορίας. Τι γίνεται τώρα. Γίνεται ότι μετά από διαβουλεύσεις που είχαμε με τους διάφορους εταίρους έχουμε τη γνωμοδότηση πια για το θέμα των αδειών των κυβερνητών και η άποψη αυτή συνάδει με τις προδιαγραφές που ισχύουν στα κράτη-μέλη και που έχουν εγκρίνει και η ΚΑΟ και η GAA. Έχουν συζητηθεί τα θέματα αυτά με εμπειρογνώμονες από την Ιάσα και από τα κράτη-μέλη ήδη από το 2010 και προβλέπονται όλα αυτά στο κείμενο το οποίο σας έχουμε στείλει και το οποίο θα ελέγξει και το Συμβούλιο τον Ιούλιο. Θα συνεχίσουμε τον Νοέμβριο και ελπίζουμε τότε να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να έχουν 4-5 μήνες για να ετοιμάσουν τα συστήματα. Αυτή είναι η θεωρία. Τώρα, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Γι' αυτό και έχουμε προβλέψει μεταβατικά μέτρα στους κανόνες, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των χωρών μελών και, των, ε, και της ε, βιομηχανίας για να ανταποκριθούν στις νέες προδιαγραφές αδειών. Η μεταβατική περίοδος είναι μέχρι τις 8 Απριλίου του 2015 και για την μετατροπή το, του συστήματος διών εφόσον δεν συνάδει τώρα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται, είναι οι non-jar compliance licenses, πάλι υπάρχει μεταβατική περίοδος μέχρι το 2014. Πιστεύουμε με, ότι με τόσο μακρές περιόδους θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μία ε, ήρεμη μετάβαση χωρίς προβλήματα. Μία πρόσκοπτη μετάβαση. Στη συνέχεια, πολύ γρήγορα, η νομοθεσία αυτή βέβαια θα είναι νομοθεσία όλων των χωρών μελών. Τώρα, κάτι άλλο στις προτάσεις είναι μια συμπληρωματική πρόταση που αναφέρεται σε προδιαγραφές υγείας, ιατρικό πιστοποιητικό. Είναι υπέρ της ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θα βοηθήσει για την είσοδο πιλότων αφού προηγουμένως έχουν περάσει από τα κατάλληλα ιατρικά τεστ χωρίς να υπάρχει υπερβολικό βάρος στις αρχές και τους διάφορους φορείς. Ιδίως για αυτή την αρχική ιατρική εξέταση από την οποία περνάνε οι κυβερνήτες και το περιεχόμενο της ιατρικής αυτής εξέτασης. Πάντω ε, περιμένουμε και τη μετάφραση από την Επιτροπή και θα είναι έτοιμη και αυτή η διάταξη σύντομα. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι σε αυτού ε, του τομεί που είναι επίμαχοι, η δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνεται πάντα από την αρχή τη ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Έπειτα θέλουμε να τηρήσουμε την αναλογικότητα και την επικουρικότητα έτσι ώστε να αντικατοπτρίσετε στις αποφάσεις μας και η πολυπλοκότητα που έχει να κάνει με τα διαφορετικά είδη σκαφών και με τις διαφορετικές διαδικασίες. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες που εφαρμόζονται από τις χώρες μέλη, κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ τον κλάδο. Βέβαια, όταν προχωράτε σε ένα τέτοιο εγχείρημα είμαστε σε διαβούλευση, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Το αποτέλεσμα είναι ότι μερικά θέματα συζητιώνται έντονα, το θέμα των αδειών των κυβερνητών από τρίτες χώρες, για δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε όμως παρόλα αυτά ότι στη διαδικασία διαβούλευσης τα τα ζητήματα και το ξέρετε και από τις απαντήσεις που δίνουμε στις ε, ερωτήσεις σας. Τα θέματα αυτά συζητιώνται πλήρως και με τον κλάδο και με τις χώρες μέλη. Πιστεύουμε ότι έχουμε καταλήξει σε μια ισόρροπη πρόταση, τροποποιώντας τόσο ίσιαν μέχρι τώρα για τις άδειε αυτές. Τώρα πάντα για το θέμα αυτό των αδειών των κυβερνητών και τις ερωτήσεις του κ. Λικατροή. Τι γίνεται με τους κυβερνήτες που αναγκάζονται να έχουν δύο διαφορετικές άδειε. Υπήρχαν επικρίσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να το ρυθμίσει. Πιστεύουμε ότι έχουμε εντολή οδηγίες από τον κανονισμό 206 να ασχοληθούμε με το θέμα των πιλότων που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν οδηγούν αεροσκάφος που έχει την έδρα του εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσει για διαδότηση. Οι Αμερικανοί τώρα που βρίσκονται στην Ευρώπη δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με τους δικούς μας τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό προσπαθούμε να το λύσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως έχουμε κάνει και με αμερικανικά προϊόντα, αεροσκάφη τα οποία ε, πετάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ιδέα της επικύρωσης, η οποία δεν χρησιμοποιείται μέχρι τώρα για τα αμερικανικά προϊόντα και προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για τις άδειε των κυβερνητών. Οι άδειε αυτές μπορούν να γίνουν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προϋποθέσεις θα προταθούν και θα συμφωνηθούν στα πλαίσια της δημερού συμφωνίας. Στην περίπτωση των ΗΠΑ αυτό σημαίνει διαπραγματεύσεις ενός παραρτήματος και με χαρά σας λέω τώρα ότι η συμφωνία ε, που προτάθηκε για την 1η Μαΐου θα προχωρήσει και με το παράρτημα. Και οι Ηνωμένε το θέλουν. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σίγουρα. Έχοντας υπόψη μας λοιπόν τι ισχύει, τι ισχύει από τις δύο πλευρές για τις συμφωνίες μας με Αμερική, Καναδά και Βραζιλία και από την άλλη μεριά έχοντας υπόψη μας το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο επίπεδο αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά τα συστήματα ασφάλειας με άλλες χώρες, Η Άσα γνωμοδότησε μετά από διαπραγματεύσεις με όλου του ενδιαφερόμενους για την αποδοχή αδειών που εκδίδονται είναι εκ μέρους τρίτων χωρών και πώς τέτοιες άδειες τριών χωρών μπορούν να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΙΚΑΟ. Αναφέρονται λοιπόν οι προδιαγραφές που αναπτύσσονται στο GAA και έτσι εμείς δεν προσπαθούμε να κάνουμε καμιά επανάσταση για αυτό το θέμα αλλά οι γενικές προϋποθέσεις για την αποδοχή αδειών τρίτων χωρών εφαρμόζουν τους κανόνες που θα έχετε εδώ τον Ιούλιο. Κάτι άλλο που έχουμε σκεφτεί για να χειριστούμε αυτό το ζήτημα μετά από συζητήσεις στη Ρυθμιστική Επιτροπή είναι να δώσουμε μια μεταβατική περίοδο για δύο χρόνια για πιλότους που πετάνε στην Ευρώπη αλλά έχουν άδειες τρίτων χωρών. Για δύο ακόμα χρόνια δηλαδή θα μπορούν μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Πιστεύουμε ότι έτσι έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να εκπονήσουμε ένα νέο σωστό σύστημα για τις άδειες βάσει των διμερών συμφωνιών ασφάλειας αεροπλοίας. Πιστεύουμε ότι σε δύο χρόνια θα έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τέλος γι' αυτό και θέλω να πιστήσω εδώ την προσοχή σας, είναι η κατάσταση όσον αφορά τον Καναδά και τη Βραζιλία. Εκεί είναι κάπως πιο περίπλοκα τα πράγματα, γιατί προτείναμε ένα αντίστοιχο σύστημα, σαν και αυτό που προτείναμε για τις Ηνωμένε Πολιτείε όσον αφορά τον Καναδά και τη Βραζιλία. Ε, συζητήθηκε χθε στην ΚΑΟ για το πώς θα χειριστούμε αυτά τα θέματα με τον Καναδά και την Βραζιλία και τις συμφωνίες με αυτές τις χώρες. Και αποφασίστηκε ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή διαδικασία, δηλαδή για νέα παραρτήματα που να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία αποδοχή αδειών. Να έχουμε νέα παραρτήματα λοιπόν στι συμφωνίες με αυτές τις χώρες. Άρα πρέπει προηγουμένω το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουν εγκρίνει μια επίσημη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και καταλαβαίνω γιατί. Θέλουν καταρχήν να υπάρξει πολιτικός έλεγχος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Υπάρχει ανησυχία για το ότι η διαδικασία είναι πολύ βαριά, δεδομένου ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Φοβούμαστε ότι δεν εξυπηρετούνται έτσι τα συμφέροντα της βιομηχανίας, η οποία θέλει να υποφεληθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα από την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών των κυβερνητών. Επίσης, φοβούμαστε ότι υπάρχει μια ανισορροπία. Δηλαδή, αλλιώς βλέπουμε τις τροποποίησεις στις συνθήκες αμοιβαία ε, αναγνώρισης των ε, κυβερνητών με άλλες περιπτώσεις αμοιβαίας αναγνώρισης. Είναι θέμα της Κορεπέρ πάντως. Ελπίζω να σας εξήγησα σωστά την κατάσταση. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, Πρόεδρε, ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά. Απάντησα σε δύο από αυτά που με ρώτησε ο κ. Ελκαντρούη, αλλά υπάρχει και το τρίτο για το cruise control στις μακρινές πτήσεις. Υπήρχαν τα EU Ops σε κανονισμό που μιλάει για αξιολόγηση είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται ήδη σήμερα. Απλώ περνάει από ένα κανονισμό και πάει σε έναν άλλο κανονισμό επειδή το έχει ζητήσει η βιομηχανία. Θεωρήσαμε ότι είναι λογικό. Ελπίζω να διευκρινίζεται έτσι. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή πέρα από την μετακίνηση του τμήματος του κανονισμού από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτά. Ο κύριο Ρίκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε δόθηκαν ορισμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα ήθελα και εγώ να θέσει. Ως προς την αμοιβαία αναγνώριση αδειών έναντι των ΙΠΑ, διότι αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αφορά 100.000 ανθρώπους περίπου ετησίως, διότι υπάρχουν προσωπικές αλλά και επαγγελματικές επιπτώσεις από ό,τι άκουσα υπάρχει λοιπόν το θέμα των Αμερικανών αδειούχων που ε, έρχονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Αν μέχρι τον Απρίλιο του 2014 δεν έχει επιληθεί το θέμα, πώς θα έχει το θέμα της επάρκειας αδειών. Και θα μπορεί να υπάρχει μία προσωρινή αδιαδότηση μέχρι την ε, τελική επίλυση του θέματος ή θα χαθεί η άδεια αν δεν επιληθεί το θέμα μέχρι τον Απρίλιο του 2014, κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό για τους πιλότους. Γνωρίζουμε ότι θα γίνει μία συζήτηση, θα υπάρχει μία συμφωνία επάρκειας αναμένοντας ε, την ε, τελική απόφαση του Απριλίου 2014. Αν όμως ε, δεν θα φτάσουμε σε μια επίλυση του ζητήματος τον Απρίλιο του 2014 θα, δοθούν, θα δοθεί περαιτέρω παράτωση. Μάισνερ. <coughs> Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τον Ντομινίκ Ρικέ. Πρόκειται κυρίως για τις άδειες χειριστών, πιλότων, που έχουν αποκτηθεί στις Ηνωμένε Πολιτείε. Που μάλιστα καμιά φορά είναι και οι κανόνες εκεί πιο απαιτητικοί και από τους ευρωπαϊκούς. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν πώς είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζονται εδώ, παροιμήν, στην Ευρώπη. Είπατε τώρα ότι είναι δυνατόν να γίνει αυτό με την Air Agreement με τις Ηνωμένε Πολιτείε για να αναγνωρίζονται οι άδειε αυτέ χειριστών χωρίς να χρειάζεται ο συγκεκριμένο χειριστή να αποκτήσει δεύτερη άδεια. Αυτό κατάλαβα, αλλά θα πρέπει να μου το εξηγήσετε. Επίσης, στη συμφωνία αυτή, η συμφωνία αυτή μάλλον, θα έπρεπε να είναι στη βάση της ισότης μεταχείρισης. Καμιά φορά όμως οι Αμερικανοί έχουν το πλεονέκτημα γιατί ε, είναι απαιτητικότεροι. Τι κάνουν οι Αμερικανοί με τις άδειε χειριστών οι οποίες έχουν αποκτηθεί στην Ευρώπη. Δεν αναγνωρίζονται εκεί. Αυτό θα σήμαινε μια έλλειψη ισορροπίας ε, διότι εμείς θέλουμε αφενός να διευκολύνουμε τα πρόσωπα εκείνα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άδεια χειριστού εδώ, εδώ αυτή που απέκτησαν στις ΗΠΑ αλλά θέλουμε βέβαια και ίση μεταχείριση. Τώρα, για Καναδά και Βραζιλία. Είπατε ότι το Συμβούλιο Υπουργών θα πρέπει να εγκρίνει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με κάποια εναρμόνιση ή κάποια συμφωνία. Υπάρχει τέτοια πρόταση ήδη. Αυτό δεν το κατανόησα καλά. Είναι συγκεκριμένο το ερώτηση λοιπόν. Υπάρχει ήδη η πρόταση αυτή. Αυτά κυρίως και τώρα για το cruise relief. Από όσο ξέρω και οι συγκυβερνήτες επιτρέπεται να χειρίζονται κυρίως για μεγάλα επιβατικά αεροσκάφη εφόσον έχουν αποδείξει στον προσωμιωτή ότι είναι ικανοί να κάνουν τους απαραίτητους χειρισμούς και για την προσγείωση και απογείωση και όχι μοναχά τον έλεγχο του αεροσκάφους σε, ε, στους εθέρες, όταν ήδη δηλαδή βρίσκεται Ε, αυτά λίγο πολύ τα ξέρω διότι ο ανιψιός μου είναι πιλότος, τώρα βέβαια έχει, ε, έχει ε, γονική άδεια, αλλά δεν έχει κάνει, έχει κάνει τις εκπαιδεύσεις αυτές. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Μένουν ανοιχτά ορισμένα ερωτήματα. Με ενδιαφέρει αφενός ο συντονισμός ή εν πάση περιπτώσει η αναγνώριση σε αυτούς τους τέσσερις εναέριου χώρους τι στάση τηρούν οι Αμερικανικές αρχές απέναντι σε Βραζιλιάνους και Καναδούς, αλλά και Ευρωπαίους, δηλαδή σε Καναδικές, Βραζιλιάνικες και Ευρωπαϊκές άδειε. Είπατε επίσης ότι με Βραζιλία και Καναδά τα πράγματα θα είναι κάπως δύσκολα. Πού εντοπίζονται οι δυσχέρειες. Είναι τα πράγματα έτσι όπως συνήθως ότι δεχόμαστε ό,τι λένε οι Αμερικανοί Πέφτουμε δηλαδή στα τέσσερα μπροστά τους και αυτοί υπαγορεύουν και διατάσσουν. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Έχω λίγο την εντύπωση, γνωρίζω και εγώ πολλούς Ευρωπαίους πιλότους οι οποίοι απέκτησαν την άδεια χειριστού στην Αμερική επειδή είναι φθηνότεροι και ευκολότεροι. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα, δηλαδή Θα ήθελα να μάθω εάν οι δικές μας εξετάσεις είναι τόσο απειρχιωμένες, είναι τόσο παραφορτωμένες, ώστε ρωτούν τους ε, χειριστές εκεί πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Θα ήθελα λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τα θέματα αυτά, διότι μέχρι τώρα δεν είναι η εικόνα πολύ καθαρή. κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. ένα θέμα ε, πληροφόρησης ε, σε σχέση με τα προγράμματα πλεύσης ε, ως προς τους κυβερνήτες και συγκυβερνήτες όταν έχουμε να κάνουμε με υπερατλαντικές πτήσεις θα πρέπει ο κάθε κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης να ε, μπορεί να αναπαύεται. Πρόκειται για μια πρακτική που ισχύει και γι' αυτό ε, υπάρχουν συγκυβερνήτες που έχουν την ίδια εκπαίδευση με τον κυβερνήτη. Άρα αυτό το θέμα δεν είναι θέμα ουσίας, όπως είπε και ο Μάθιου Μπόλτουιν. Απλώς μεταφέρονται τα ίδια ε, δεδομένα και ισχύουν και στην περίπτωση του ενός και του άλλου. Είναι πολύ καλό το ότι είχαμε αυτή τη συζήτηση, διότι αυτό που έχει σημασία είναι η αδειοδότηση τρίτων χωρών από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών στην Ευρώπη υπήρχε αμοιβαία αναγνώριση αυτών των αδειών διαχρονικά. Δεν είναι σοβαρό το ζήτημα οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θεώρησε ότι αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι στις ΗΠΑ είναι πολύ καλοί πιλότοι, δεν ετέθησαν θέματα ασφαλείας. Πολλοί εργάζονται στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το χρονοδιάγραμμα του 2014 Υπάρχουν πολλοί προσωμιωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν ε, βεβαίως οι εκπαιδευτές και θα πρέπει να τους λάβουμε και αυτούς υπόψη. Η διατύπωση είναι λίγο διαφορετική εδώ. Ενώ μιλούσαμε για Ευρωπαίους πολίτες, μιλάμε για ε, κατοίκους, εκείνους που διαμένουν στην Ευρώπη. Μιλάμε όχι πια για citizens, αλλά για residents. Δεν θα θέλαμε να έχουμε χιλιάδες ε, πιλότους που να εργάζονται στην Ευρώπη και που ξαφνικά να μην έχουν εργασία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εάν θα πρέπει να κινηθούμε από τη μία άδεια στην άλλη, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση. Εάν Υπάρχουν ε, πιλότοι στην, στη ΣΥΠΑ που μπορούν να εργαστούν στη ΣΥΠΑ θα πρέπει να μπορούν να εργαστούν να πούμε ότι δεν υπάρχει σωστή εκπαίδευση ή ότι δεν υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας. Θα πρέπει να μιλήσουμε ως ενήλικες. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα παραρτήματα και ο Μάθιου Μπόλντουιν το, το τόνισε αυτό. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε ε, ένα απλουστευμένο σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση καταλογικό τρόπο. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε κυρώσεις ε, κατά τον μεν ή τον δε όταν μιλάμε για υποχρεωτικές 150 ώρες γιατί υπάρχουν πολύ, υπάρχουν πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Εγώ δεν, ως επιβάτης δεν ε, ασχολούμαι με το κατά πόσο ένας πιλότος που με μεταφέρει στην Αμερική ή στην Ευρώπη έχει άδεια ευρωπαϊκή ή αμερικανική. Ελπίζω η Κομισιόν και η Άσα να φτάσουν σε ένα λογικό συμβιβασμό έτσι ώστε να έχουμε μια καλή μετάβαση στους κοινούς κανόνες αεροπλοείας. Αυτό είναι το θέμα ουσίας. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τα σχόλιά της. Ο κύριος Μπράντμπορν. Ευχαριστώ. Γενικά θα ήθελα να θίξω το εξής με προσέγγισαν πολύ στην εκλογική μου περιφέρεια. Ιδιαίτερα για τις ε, πτήσεις αναψυχής, όπως τις αποκαλούμε. Και από όσο γνωρίζω, υπάρχουν, ε, υπάρχει πρόβλημα να εισακουστούν αυτοί οι άνθρωποι γιατί η Επιτροπή η ΆΣΑ δεν κοινοποιεί αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αποτανθούν στην ασα Δεν υπάρχει διαφάνεια. Η Κομισιόν θα θέλει να προβάλλει μια καλύτερη εικόνα. Γιατί, πρέπει γιατί δεν πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα και να υπάρχουν απόρριτα δεδομένα. Κάθε φορά που έρχομαι σε αυτή την επιτροπή μιλάμε για κάποια αποτυχία με βάση την ε, λήψη απόφασης, μια λήψη απόφασης σε επίπεδο η Ο Πίτερ Παντόλεν μας ε, έκανε μια πολύ καλή ενημέρωση σε σχέση με τις αντιρρήσεις του ως προς αυτό το έγγραφο, ως προς τον ε, τομέα πολιτικής αεροπλοείας. Θα ήθελα να θίξω ορισμένα ζητήματα που με ανησυχούν ιδιαίτερα. Πρώτον, αυτή η απόφαση της ΙΑΣΑ απειλεί ένα σύστημα το οποίο ήταν αποδεκτό διεθνώς ανά τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μία λύση χωρίς να υφίσταται πρόβλημα, για να το θέσω έτσι. Η κατοικία των πιλότων δεν έχει καμία σημασία διότι σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις οι πιλότοι που μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή άδεια ανεξάρτητα από το που, ποια είναι η έδρα της αεροπλοείας. Αυτό όμως θίγει τους Ευρωπαίους πιλότους με ευρωπαϊκή άδεια, διότι στις ΗΠΑ μπορούμε να έχουμε πιλότους οι οποίοι έχουν πάρει άδεια στην στις ΗΠΑ, αλλά μπορούν να διαμένουν στην Ευρώπη. Ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο. Αυτό είναι ένα παράλογο σύστημα αντιπαράθεσης. Προβάλλουμε αυτά τα επιχειρήματα περί ασφάλειας και ούτω καθεξής, μα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτές οι άδειες, οι δικές μας, οι ευρωπαϊκές, δεν πληρούν τα εχέγγυα ασφάλειας. Υπάρχει μαύρος κατάλογος και στην ε, Ευρώπη, όπως υπάρχει και στις ΗΠΑ. Το θέμα είναι το κόστος, δεν είναι ίσονος σημασίας. Εάν πρέπει να γίνει μετατροπή, γιατί μιλάμε για 68.000 πιλότους που είναι εμπλεκόμενοι, τότε το κόστος συντηρητικά, το κόστος επανεκπαίδευσης εκπαίδευσης είναι 120 εκατομμύρια λίρες. Άρα δεν είναι αμεληταίο το ποσό. Έχουμε αεροπλάνα, ε, μάλλον ε, αερο, εταιρείες οι οποίες δεν θα έχουν πρόβλημα με τη ΣΥΠΑ διότι θα υπάρξουν άλλες συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ. Αυτό όμως σημαίνει επιμερισμός σημαίνει επιμερισμό. Όταν θα λάβουμε την πρόταση τον Ιούλιο, όπως μας ελέγχθη, θα πρέπει ως Κοινοβούλιο να ε, απορρίψουμε αυτή την πρόταση μέχρι ότου φτάσουμε στην επίλυση του ζητήματος έτσι ώστε αυτοί που έχουν αμερικανικές ε, άδειες να μην ε, έχουν διακρίσεις, γνωρίσουν διακρίσεις επειδή διαμένουν στην Ευρώπη. Πρόεδρος, δεν θα μιλούσα, α, αλλά κύριε Μπράντμπον, εγώ δαπανώ μεγαλύτερο χρόνο λόγω αποτυχίας διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και όχι με την Ιάσα, μιλώντας για αποτυχίες. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο πέρασε τον κανονισμό 216 που μιλά για ευρωπαϊκές άδειες μετά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε ευρωπαϊκές άδειες γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα. Το συμφωνήσαμε το 2008 ότι αυτό θέλαμε και ο κύριος Αλκαντράου έχει δίκιο όταν είπε εξ αρχής ότι αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή θέλουμε άδειες, ευρωπαϊκές άδειες, όχι εθνικές. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης. Η κυρία Φώστερ έχει δίκιο όταν μιλάει για συγκυβερνήτες. Όταν ε, ε, μιλά ε, για ε, τους πιλότους, τους συγκυβερνήτες, κατά πόσο θα είναι περισσότεροι ή όχι. Μπορεί κανείς να πετάξει εντός είπα με ένα συγκυβερνήτη ο οποίος δεν έχει άδεια για το συγκεκριμένο αεροσκάφος ορισμένοι αμερικανικοί κανόνες δεν είναι και τόσο σωστοί. Ο συγκυβερνήτης ε, κυβερνά ένα αεροπλάνο για το οποίο δεν έχει άδεια. Άρα η κυρία Φώστερ έχει δίκιο όταν μιλά για το, θέμα ενισχυμένου, ε, ενισχυμένου σχήματος πιλότων και συγκυβερνητών. Κύριε Μπόλτιν, να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, αλλά μιλάμε για αμοιβαία αναγνώριση αδειών. Και είπα, δεν αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές άδειες πιλότων. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο και αν λάβω υπόψη αυτά που είπε ο κύριος Μπράτμπορν, θεωρώ ότι οι αμερικανικές άδειες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή οι ευρωπαϊκές άδειες να γίνονται αποδεκτές της ΕΠΑ. Άρα, εάν οι ΕΠΑ δεν τις αναγνωρίζουν, γιατί πρέπει εμείς να αναγνωρίσουμε τις δικές τους άδειες, γιατί να αναγνωρίσουμε τις αμερικανικές άδειες. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ το τόνισε. Δηλαδή μας υποδεικνύουν και πάλι είπα τι θα πρέπει να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ε, στην ουσία αποδεχόμαστε τους όρους ε, αμελητή. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ε, με μια αμερικανική άδεια, αλλά και οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να έχουν πρόβλημα με τις δικές μας άδειες. Μέχρι το 2014 θα πρέπει να επιλύσουμε το θέμα. Ίσως όμως θα ήταν σκόπιμο να ασκήσουμε πίεση προς τη ΣΥΠΑ, όπως έκανα και εκείνη έναντι της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να είμαστε ίσοι. Άρα, κύριε Πόλτουιν, υπάρχουν αυτά τα δύο χρόνια για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία με τις ΙΠΑ. αλλά εγώ είμαι ειλικρινής. Ειλικρινής, αν δεν ε, είναι σωστό το παιχνίδι των ΙΠΑ, δεν θα πρέπει να είναι ούτε και το δικό μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς πρέπει να υποχρούμε συνέχεια. Αλκαντράουι, η Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει Νομίζω ότι οι συνάδελφοι ενίσχυσαν τις δικές μου ερωτήσεις. Ας απαντήσει η Κομισιόν και μετά θα δούμε τι θα κάνουν. Εντάχει παρακαλώ. Ε, ξέχασα. Γιατί υπάρχει και το θέμα της ηλικίας, της διάκρισης με βάση, των διακρίσεων με βάση την ηλικία υπάρχει ε, ε, διάκριση ως προς την ηλικία σε σχέση με τις ε, ιατρικές εξετάσεις. Ίσως όχι, αλλά θα δούμε. Και μας μας δυσκολεύει αυτό. Ελπίζω να έχουμε βρει την απάντηση μέχρι να τελειώσω. Το ψάχνουμε. Με τη σειρά θα απαντήσω. Ήταν πολύ χρήσιμες οι ερωτήσεις. Στον κύριο Ρίκε πρώτα να απαντήσω. Η δικιά σας ανησυχία, κύριε Ρίκε, ήταν ότι θα υπάρξει κενό αν δεν μπορέσουμε μέσα στα δύο αυτά χρόνια να έχουμε διαπραγματευτεί. Θα έχουμε εξαντλήσει το χρόνο. Αυτό που συμφωνήσαμε, και έχετε δίκιο, ε? και επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος, δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε βάσει του ότι α, δεν έχουμε χρόνο, γιατί τότε είναι που δεν είναι καλές διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται να έχουμε ελαστικότητα όσον αφορά το χρόνο. Λοιπόν, αυτό που συμφωνήσαμε είναι ότι η απόφαση για τη μεταβατική περίοδο θα είναι κάτι που θα ελέγξουμε εμείς. Και οι διαπραγματεύσεις θα μπορέσουν να ελεγχθούν σχετικά εύκολα. Τώρα, όταν θα περάσει ο χρόνο, θα δούμε. Χρειάζεται να παραταθεί μεταβατική περίοδος. Δεν θέλω να προκαταλάβω καμία απόφαση, αλλά λογικό θα ήταν ε, μετά από αυτά που είπατε για το κόστος, τις δυσκολίε και ε, τις δυσκολίε που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος. Θα δούμε τότε τι θα κάνουμε. Δεν θέλουμε δηλαδή να βρεθούμε τον Απρίλιο του 2014 ε, κολλημένοι στον τοίχο χωρίς να έχουμε καμία διέξοδο. Για την κυρία Μάισνερ. Οι ερωτήσει για την ασφάλεια και για αυτά που είπε ο κύριος Μπάλτουιν το λέω. Μία από τις ανησυχίες που είχαμε και που συμμεριζόταν και το Κοινοβούλιο το 2008 όταν μας έδωσε την εντολή είναι ότι δεν υπήρξε πάντα δυνατότητα εφαρμογής απέναντι σε κυβερνήτες τρίτων χωρών. Και αυτό είναι που θέλουμε να ξεπεράσουμε για να έχουμε ασφάλεια. Έπειτα, η αντιστοιχεία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό είναι κάτι που είναι η κόκκινη γραμμή για μας και συμφωνούμε. Οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι μονόπλευρες. Αν δεν έχουμε αναγνώριση των δικών μας αδειών από τις Ηνωμένε πολιτείες, προφανώς ούτε θα αναγνωρίζονται δικές του άδειε. Και τι χρειάζεται για να το αποφύγουμε αυτό είναι διαπραγματεύσεις ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και των δύο πλευρών, να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια και να καθισχάσονται και οι δύο πλευρές. Τώρα, για το cruise relief, αυτό που είπε και η κυρία Φώστερ, στην κατάσταση που περιγράφεται όταν έχουν λείψει για καιρό, πρέπει να απαιτούνται από αυτούς, να απαιτείται από αυτούς ε, κατάρτιση, πρόσφατη κατάρτιση. Κυρία Λίχτεμπέργκερ, ίσως να μην ήμουν αρκετά σαφής στην αρχή. Όταν είπα ότι τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα και ίσως πιο δύσκολα για τον Καναδά και την Βραζιλία, αναφερόμουν στις διαδικασίες όταν θα διαπραγματευτούμε τα νέα παραρτήματα. Φυσικά δεν θέλω εδώ να μιλήσω εκ μέρους του Συμβουλίου, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω τι κατάλαβα ότι συμφώνησαν χτες στο Συμβούλιο και Κορεπέρ. Και αυτό ήταν πλήρης ευρωπαϊκή διαδικασία για εντολή της ε, κοινή Επιτροπής να συμφωνήσει για νέα παραρτήματα. Χρειάζεται συμφωνία της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τις προτάσεις. Δεν γίνεται βάση απόφασης του Συμβουλίου γρήγορα και τίποτα άλλο. Δεν προσπαθώ να ε, φέρουν αντιρρήσει στην ε, πρόθεση του Συμβουλίου να προχωρήσει σε εποπτεία των κανόνων όπως θέλει. Απλώς αυτό δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στη βιομηχανία εν ώψη των συμφωνιών αυτών με τον Καναδά και την Βραζιλία. Πάντως ευχαριστώ την κυρία Φώστερ για αυτό που είπε. Για το πόσο ευαίσθητα είναι τα ζητήματα. Πράγματι φάνηκε αυτό και σήμερα. Έτσι κι αλλιώς, κύριος στόχος μας είναι η ασφάλεια και η σωστή εφαρμογή των κανόνων. Τώρα, στα θέματα του κύριου Μπάλτουιν. Και ευχαριστώ. Κύριο Μπράντμπορτ. Αναφερθήκατε στις ε, ομάδες ενδιαφερόντων που μερικές φορές δυσκολεύονται όταν έχουν δύσκολη πρόσβαση για να φτιάξουν ε, τους κινητήρες, για παράδειγμα. Η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες να μπορούν να συναντηθούν με την Brussels Sport Association και καταλαβαίνω ότι πάντα υπάρχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και όσον αφορά και την πρόσβαση στην Ιάσα. Η Επιτροπή, η ΙΑΣΑ, οι εκπροσωπή δηλαδή. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση από την κυρία Λίντεμπεργκερ, να σταματήσω, Πρόεδρε. Ευχαρίστω να σας ακούσω μετά. Έχοντας ακούσει όλα τα επιχειρήματα, τα κρατημέλη, η Άσα, η Επιτροπή, μετά θα αποφασίσουν. Πάντως τον έλεγχο το κάνει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεν είναι η Επιτροπή μόνο. Έχοντας ακούσει και την Ιάσα και άλλες επιτροπές Για την ουσία τώρα τον όσο είπε ο κύριος Πρότπορτ. Και έχω και ένα σημείο μου από τον κύριο Βαντάλεν. Θα απαντήσω. Όπως τόνισε και ο Πρόεδρος, συμφωνήθηκε από το Κοινοβούλιο ότι θέλουμε ευρωπαϊκές άδειες. Αυτό αποφασίστηκε το 2008. Τώρα δεν θέλω να βασιστώ μόνο σε αυτό το επιχείρημα, στο δηλαδή «Ε, αφού το αποφασίσαμε τελεία και παύλα. Όχι, πιστεύουμε όντω ότι είναι καλό. Και αν μπορούμε να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικά στα πλαίσια της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχουμε μία κατάσταση όπου θα υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση αδειών από τις δύο πλευρές. Τα σενάρια τρόμου, στα οποία αναφερθήκατε, ε, θα εξεταστούν αν έχουν αποτύχει διαπραγματεύσεις. Αυτό ισχύει και για το θέμα του κόστους, που αναγνωρίζω ότι είναι και αυτό ένα πρόβλημα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Ένα ικανοποιητικό επίπεδο ε, ισότητας μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν μπορούμε πάντα να διασφαλίσουμε την αποδοχή και την εφαρμογή των δικών μας προδιαγραφών, Πάντως πιστεύουμε ότι κάποιες από τις αμερικανικές άδειες όντως πρέπει να συμμορφώνονται με επιπλέον προδιαγραφές και απαιτήσει. Η Συμφωνία Ασφάλειας είναι πάντως η σωστή βάση πάνω στην οποία πρέπει να διαπραγματευτούμε. Τέλος, δεν προσπαθούμε να έχουμε καμία επανάσταση στους κανόνες, αλλά βασιζόμαστε στην αρχή της μεταφοράς των ε, διατάξεων, δηλαδή δεν αλλάζουν. Αν τα καταφέρουμε και θα φροντίσουμε να γίνει αυτό με τις διαπραγματεύσεις, αν τα καταφέρουμε λοιπόν τόσο το καλύτερο. Έτσι καλώς και οι Αμερικανοί θέλουν να προχωρήσουν με τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζουμε ότι θα έχουν καθησυχαστεί έτσι οι ανησυχίες σας το τελευταίο που μας ρωτήσατε τώρα, που έχει να κάνει με τις ιατρικές εξετάσεις και τις απαιτήσει σχετικά με τη συχνότητα των ιατρικών εξετάσεων. Μας ρωτήσατε για διακρίσεις βάση ηλικίας. Υπάρχουν οι άδειες για τα καφέ αεροσκάφη. Δεν υπάρχει όμως διάκριση βάση ηλικία στην ρύθμιση στην οποία εσείς αναφέρεστε. Όχι. Σίγουρα πολλά είναι λεπτά τεχνικά ζητήματα και άλλα είναι λεπτά πολιτικά ζητήματα. Ό,τι άλλες ερωτήσεις έχετε είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Το θέμα της ηλικίας απαντήθηκε. Όχι, δεν απαντήθηκε ως προς την αποδοχή ε, αδειών από τον Καναδά, τη Βραζιλία και την Ευρώπη. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσο είναι αναγνωρισμένες αυτές οι άδειες. Οι Βραζιλιάνοι έχουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς αυτή τη στιγμή, κύριε Μπόλτουιν οι ευρωπαϊκές άδειες δεν είναι αποδεκτές και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Από όσο ξέρω, η Βραζιλία επίσης δεν έχει την ίδια επάρκεια επάρκεια η αναγνώριση της ΕΠΑ. Θα ήθελα όμως να το ελέγξω. Για τους Καναδούς ε, δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση. Μπορείτε να απαντήσετε στην κυρία Λίχτενμπέργκερ Ναι, έχετε το λόγο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Μπόλτουιν, το εξής. Μιλήσατε για μία πρόταση της Κομισιόν που θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο σε σχέση με τις άδειε από τον Καναδά και τη Βραζιλία. Υπάρχει αυτή η πρόταση επιτάπητος ή θα συμβεί από όσο κατάλαβα προγραμματίζεται. Υπάρχει όμως ή ακόμα όχι. Κύριε Μπόλτουιν. Ε, μου είπατε ότι δεν μπορώ να συμβουλεύω με τους ε, υπαλλήλους. Αυτό ακριβώς κάνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συζητήθηκε στην Κορεπέρ είναι να δούμε πώς θα έχει το σχήμα λήψης αποφάσεων. Και εξήγησα ε, ευγενικά τις, επεξήγησα ευγενικά τις ανησυχίες του Συμβουλίου. Κύριε Αλκαντράουι, θέλετε να πείτε κάτι... Να τα σκεφτούμε όλα αυτά που ακούσαμε. Και μετά θα δούμε με την Επιτροπή τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις που έδωσε. Τίποτα άλλο. Να υπενθυμίσω στους βρουλευτές ότι η διαδικασία είναι η διαδικασία ελέγχου. Έχουμε δικαίωμα άρνηση κυρίας. Προ το παρόν δεν υπάρχει σε όλε τι γλώσσε μεταφρασμένο το μέτρο. Όταν θα έχει έρθει στο Κοινοβούλιο σε όλε τι επίσημε γλώσσε, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρει μήνε στη διάθεσή του για να ε, φέρει αντιρρήσει. Και βάσει του κανονισμού, ο πρόεδρο θα θέσει προθεσμία προκειμένου οι ευρωβουλευτέ ε, να προτείνουν ότι αντιρρήσεις έχουν. Αν γίνει αποδεχτή η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σας υπενθυμίζω ότι είναι η Επιτροπή Μεταφορών που παίρνει την απόφαση, όχι ολομέλεια. Τέλη Μαΐου ξεκινάει η περίοδος συζήτησης με τα άλλα θεσμικά όργανα. Οπότε προκειμένου να τηρήσουμε τα η περίοδος για αντιρρήσεις θα ξεκινήσει τελικά από τον Ιούλιο ώστε η πρόταση για αντίρρηση με σχέδιο ψηφίσματος θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Μεταφορών τον Σεπτέμβριο. Εντάξει. Στα διάφορα. Κύριε Μπάλτουιν, η τέφρα το... Πώς πάει... Δεν ξέρω το όνομα αν είναι πιο εύκολο φέτος, γιατί πολλοί είχαμε μεγάλη δυσκολία να προφέρουμε το όνομα του περσινού ηφαιστείου. Το ήξερα το όνομα, αλλά το ξέχασα. Grimms κάπως έτσι. Πάντως θα ασκηθώ και την επόμενη φορά θα το προφέρω τέλεια. Είπατε σε προηγούμενη συζήτηση ότι ίσως χρειαζόμαστε και άλλα ηφαίστεια για να λειτουργήσει επιτέλους ο νέος Ευρωπαϊκός Ουρανός. Αυτή η φράση σας μου προκάλεσε σκέψεις και θυμήθηκα το περίφημο «Μιλάει στο Βιετνάμ» που είχαν πει τότε οι Αμερικανοί στρατιώτες ότι χρειάστηκε να καταστρέψουμε το χωριό για να το σώσουμε. Συνεχίστε να φωτίζετε το θέμα με αυτόν τον τρόπο κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο για όλους μας να βρισκόμαστε σε παρόμοια κατάσταση όπως αυτή που ε, είχε σημειωθεί πέρσι ή ε, φαίνεται να πάει προς τα και φέτος. Εμείς οι τεχνοκράτες πρέπει να σκεφτόμαστε καμιά φορά και τις επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, τις επιχειρήσεις τους κλπ. Διακόπτη και ιδίως για την πτήση Βρυξελών-Μάντσεστερ ή και Λίβερπουλ. Ας αφήσουμε τα αστεία ωστόσο μας κρατούν όμοιρο οι μετεωρολογικές συνθήκες. Μου λένε οι μετεωρολόγοι ότι φέτος τα πράγματα είναι πολύ λιγότερο σταθερά, διότι πέρσι το σύννεφο είχε εγκατασταθεί μονιμότερα πάνω από τον ευρωπαϊκό Ενέριο χώρο. Τώρα έχουμε ένα άλλο σύστημα μετεωρολογικό, δηλαδή με ψυχρά μέτωπα τα οποία έρχεται είναι δύσκολο να κάνουν πρόγνωση για τις επόμενες 4-5 ημέρες. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι πέρσι. Γι' αυτό η Ευρωκοντρόλ κάνει τακτικές ενημερώσεις και δεν προσπαθεί, δηλαδή καθημερινές, και δεν προσπαθεί να προβλέψει για 36 ώρες. Θα είδατε επίσης ότι η τέφρα έχει διαφορετική, ε, διαφορετικό ποιόν. Θα πέσει λοιπόν στο έδαφο ταχύτερα. Είναι διαφορετική και η έκρηξη και ίσως ενδεχομένως και η διάρκεια της ίσως ήδη είχε αρχίσει να μειώνεται η ισχύ της. Όλα πάντως αυτά κάνουν δυσκολότερο να γίνουν προβλέψεις. Ένα πράγμα που ωστόσο δεν άλλαξε, για να το πω ειλικρινά, είναι ότι ο ενέργειος χώρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κυριαρχία των χωρών μελών. Και το εάν θα ανοίξει ή θα κλείσει ο ενέργειος χώρος είναι υπόθεση της συγκεκριμένης χώρας μέλους. Ε, προσπάθησα και πριν να το πω αυτό όταν συζητούσαμε τα λεγόμενα Functional Airspace Block, τα FAB. Μιλούμε ωστόσο για ένα δίκτυο, ένα δίκτυο του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου. Και περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα ευεργετήματά του. Υπάρχουν δύο μεγάλες διαφορές φέτος. Ήδη από σήμερα, ήδη μάλλον λειτουργεί η Επιτροπή Κρίσης που στην ουσία ε, με τηλεφωνικές συνδιαλέξεις καθημερινά και συνδιασκέψεις ε, παρακολουθούμε καθημερινά και πολύ τακτικά την κατάσταση. Έτσι λοιπόν υπάρχουν... Α, κλείνει το μικρόφωνο του. Με συμμετοχή όλων των ε, συνδικάτων των ελεγκτών αέρια κυκλοφορίας, όλων των υπευθύνων, με πολύ σφιχτή ατζέντα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, διατηρήσουμε τα υψηλά επίπεδα ασφάλεια χωρίς να κλείσουμε συνολικά τον ενιαίο χώρο. Το άλλο θέμα είναι ότι έχουμε και τις κατευθύνσεις γραμμέ τη ΙΚΑΟ που λειτουργούν και που δείχνουν πώς, και μας εξηγούν πώ μπορούμε να κάνουμε safety risk assessments από τις ε, ε, εταιρείε σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές για να επιτρέψουν στις εταιρείε με πάρα πολύ στοχευμένο τρόπο να εξετάσουν εάν είναι ασφαλές να πετάξουν τα αεροσκάφη τους και να λάβουν και την έγκριση από τις εποπτικές αρχές. Οι κεντρικές αρχές, ωστόσο, αυτό σημαίνει είτε στη χώρα μέλος είτε από τη σκοπιά του Ευρωκοντρόλ δεν θα είναι, να μην είναι δηλαδή ανάγκη να πούν «Α, πρέπει να κλείσουμε αυτό τον αέριο χώρο». Και αν δούμε τι είναι στις 24 τελευταίες ώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, χάσαμε 250 πτήσεις που ακυρώθηκαν δηλαδή, το οποίο βεβαίως δυσκολεύει τη ζωή αυτών που θα πετούσαν με αυτά τα αεροσκάφη, αλλά τουλάχιστον δεν ανέβηκαν ε, οι αριθμοί σε χιλιάδες ε, πτήσεις. Η πιο πρόσφατη περιγραφή της καταστάσεως είναι ότι οι, όλες οι χώρες μέλη εφαρμόζουν την προσέγγιση SRA και ορισμένα τμήματα του γερμανικού εναέριου χώρου είναι κλειστά πάνω από την Πρέμη και το Αμβούργο σε σχετικά χαμηλότερα ύψη και γύρω από το Βερολίνο. Η κατάσταση στο Ενωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι θα χαλαρώσει μέσα στη σημερινή ημέρα. Βέβαια ακόμα ορισμένα αεροσκάφη έχουν μείνει αλλού από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Έγινε πάλι η σύσκεψη σήμερα και είμαι βέβαιος κύριε Πρόεδρε ότι έχουμε δει διαφορές προσέγγισης από διάφορες χώρες μέλη στο θέμα της κρίσης αυτής. Βέβαια το κλείσιμο του ενέργειου χώρου στην ε, Γερμανία σήμερα έχει γίνει πολύ στοχευμένα γύρω από τη Βρέμη και το Αμβούργο όπως είπα και οι πρακτικές επιπτώσεις, οι επιπτώσεις στην πράξη δηλαδή, θα είναι σχετικά περιορισμένες. Θα ήταν χρήσιμο να προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε μέσω ημών ή μέσω της γραμματείας αν μπορούμε μάλιστα και γραπτός να σας ενημερώνουμε γραπτός αυτό νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο γιατί βεβαίω και οι πολίτες θα στραφούν σε εσά για να σας ερωτήσουν ευχαριστώ κύριε Μπόλτιν μπορείτε να τα διαβάσετε σε μένα και εγώ πολύ ευχαρίστω θα τα διαβάσω σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέλος της Επιτροπής Μεταφόρων Ευχαριστώ. Έχετε ερωτήσεις αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε ευγνώμονες για την ενημέρωση. Ελπίζω αυτό το συγκεκριμένο εφέστιο να σιγήσει και πάλι γρήγορα και να επανέλθουμε σε φυσιολογικά όρια. Άλλος κανείς έχει κάτι στα διάφορα. Εάν όχι... Να ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς και